Proszę Państwa, prawie Με καθυστέρηση περίπου 15 λεπτών ξεκινάμε. Ε, θα συνεδριάσουμε σε τρεις ε, ενότητες σήμερα το απόγευμα, αύριο το πρωί και αύριο το απόγευμα. Αν δεν υπάρχει παρατήρηση μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και πληροφοριακά μπορώ να σας πω και θέλω να σας πω ότι ε, υπάρχει διερμηνία, μεταδίδεται διερμηνία μέσω ε, διαδικτύου. Εκτός από μαλτέζικα, σλοβάκικα και ε, κέλτικα, όλες οι άλλες γλώσσες υπάρχουν στη συνάντησή μας σε ταυτόχρονη διερμηνία. Έχουμε λοιπόν τα πρακτικά που σας έχουν κατατεθεί. Η κυρία Πόλσεν θα ξεκινήσει με το σημείο υπαριθμών 4. Ο κύριος Μπούλα πρέπει να φύγει και η κυρία Αγκουλιέρα η οποία είναι εισηγήτρια στο πέμπτο σημείο Παρασκευή διάθεση στα αγορά και χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών και καταρτιση της οδηγίας 90-167 όκτου Συμβουλίου ε, θα προηγηθεί. Επ' αυτού έχουν συμφωνήσει δύο κυρίες ε, ε, να κάνουν σκάτζερ, το 5 να γίνει 4 και το 4-5. Αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Γεωργίας. Ε, γνωμοδότηση θα πάρουμε από την Επιτροπή ε, περιβάλλοντος. Δεν θα κάνω εισαγωγή επί του θέματος. Η κυρία Αγγιλέρα ε, είναι πιο κατάλληλη για να κάνει την εισαγωγή της έκθεσής της και θα μας παρουσιάσει αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που είναι η παρασκευή διάθεση στην αγορά και χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών. Υπάρχουν και πολλά άλλα παρεμφερή θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Πρόκειται για τα φάρμακα. Πρόκειται γενικότερα για την υγεία των ζώων. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα ήθελα να σας δώσω το λόγο, ε, κυρία εισηγήτρια, ε, Προηγούμενο όμως επιτρέψτε μου να καλωσορίσω πολλονούς φοιτητές ε, οι οποίοι ασχολούνται με αυτόν τον τομέα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας καλωσορίζω όλους θερμά. Είμαστε όλοι στη διάθεσή σας, κυρίως εγώ. Αν έχετε ερωτήσεις μπορείτε να τις υποβάλλετε μετά τη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής. Και παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο. Bueno, buenas tardes. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Να καλωσορίσω και τους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες μας και είμαστε στη διάθεσή τους φυσικά, όπως είπε και ο Πρόεδρος, για οτιδήποτε χρειαστούν. Δεν ξέρω κύριε Πρόεδρε τι χρόνο έχω στη διάθεσή μου για να σας παρουσιάσω την έκθεση. Εντάξει. Θα είμαι συνετή ε, στο χρόνο αγόρευσης. Θα σας μιλήσω λοιπόν για την έκθεση μου της προτάσεως κανονισμού για τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Αρμόδια καθήλυν είναι η Επιτροπή μας, το είπε και ο Πρόεδρος, όμως σχετίζεται με άλλους δύο κανονισμούς. Ε, ο ένας αφορά τα κτηνιατρικά φάρμακα και το δεύτερο το νέο οργανισμό για κτηνιατρικά θέματα. Θέλω να πω ευθύς εξ αρχής και είναι σημαντικό αυτό. Κάποιο πρόβλημα υπήρχε με τη διερμηνία από τα ισπανικά προς τα γερμανικά. Εντάξει τώρα. Bueno, el Μάλιστα, ωραία. Λύθηκε το ζήτημα αυτό, το γλωσσικό και συνεχίζω. Έλεγα λοιπόν ότι ναι, μεν εμείς είμαστε καθήλυνα αρμόδιοι ως Επιτροπή για αυτό τον πολύ σημαντικό κανονισμό Είπα ότι η σημαντική, κατά την άποψή μου, αλλά και κατά την άποψη των συνάδελφων την οποία γνωρίζω, το κ. Λίν, ότι είναι σημαντικό ο κανονισμός αυτός χρονικά να εξεταστεί στο ίδιο χρονοδιάγραμμα με τον βασικό κανονισμό για τα κτηνατικά φάρμακα. Γιατί υπάρχουν ζητήματα που αφορούν και τον ένα και τον άλλο κανονισμό Άρα δεν είναι λογικό να προχωρήσουμε με έγκριση ενός ε, κανονισμού πολύ πιο γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν εντάξαμε στο ίδιο χρονοδιάγραμμα τους δύο κανονισμούς, τις ε, δύο εκθέσεις. Φαντάζομαι ότι έχετε διαβάσει τον, την έκθεση, αλλά θα σας παρουσιάσω και τα βασικά της ε, σημεία και είμαι και στη διάθεσή σας βέβαια οι οτροφέ είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ομάδων ζώων, όχι με μονομένα ζώα δηλαδή, αλλά έχουν ακριβώς ένα βαθμό αποτελεσματικότητας ό,τι αφορά ομάδες ζώων. Και κατά την άποψή με τον τρόπο αυτό εγγυούμεθα μια πιο ομοιογενή και σταθερή κατανομή. Κάθε ζώο λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο έχει πρόσβαση σε ίδιες ποσότητες ε, φαρμάκου μέσω αυτής της φαρμακούχα ζωοτροφής και στην ενδεδειγμένη ποσότητα που απαιτείται ώστε να είναι ώστε να τον πιο αποτελεσματική αγωγή. Φυσικά άποψή μου είναι αυτή, αλλά θέλω να σας το πω ευθύς εξ αρχής. Δηλαδή, ομάδες ζώων, όχι μεμονωμένα ζώα, και είναι πιο ομοιογενής η θεραπεία, άρα και πιο αποτελεσματική στην προκειμένη περίπτωση. Πρέπει να σας πω επίσης ότι οι φαρμακούχες ζωοτροφές είναι μία μόνο από τις πολλές θεραπευτικές εναλλακτικέ για την αποτουστώματος χορήγηση του κτηνιατρικού φάρμακου αμαδεζών. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, τα διαλυτά φάρμακα, δηλαδή ανάμεξη πόσων νερού με κτηνιατρικά φάρμακα ή όταν ο κτηνοτρόφος διανέμει με το χέρι τα φάρμακα αυτά, κάποια ουσία πάνω στη ζωοτροφή. Άρα οι φαρμακολογικές ζωοτροφές είναι μία ακόμη εναλλακτική. Κατά την άποψή μου, προσφέρει μεγαλύτερη ομοιογένεια αυτή η εναλλακτική. Αλλά είναι μία εναλλακτική θεραπευτική αντιμετώπιση, μαζί με άλλες. Επίσης, οι φαρμακούχες ζωοτροφές πέραν από τους συγκεκριμένους κανόνες της οδηγίας, αν εγκριθεί ο κανονισμός, θα υπόκεινται σε αυτούς τους κανόνες. Αλλά και στη γενική νομοθεσία για τη σήμανση και την υγιεινή των ζωοτροφών καθώς και στους κανόνες για τη διάθεση στην αγορά και για τη χρήση ζωοτροφών και προσθέτων ζωοτροφών. Στο νέο κανόνισμα για τα κτηνιατρικά φάρμακα καθορίζονται βασικοί κανόνες για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Κάποια από τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακούχων ζωοτροφών. Επομένως, η επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την ορθή χρήση των ιατρικών φαρμάκων θα πρέπει να εμπίπτει κατά την άποψή μου στο πλαίσιο του λόγου κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Κατά συνέπεια η πρόταση για τις φαρμακούχες ζωοτροφές, όπως είπα και στην αρχή, θα πρέπει να εξεταστεί. Παράλληλα, ίσως λίγο, σε κάπως μεταγενέστερο στάδιο, με την πρόταση κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Αυτό το σχέδιο κανονισμού για τις αρμακούγες τροφές επικαιροποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που χρονολογείται από, το, από τη δεκαετία του 90. Ξέρω ότι έχουμε αποκτήσει εμπειρία και έχουμε περάσει και χρόνια, αλλά συνειδητοποιούμε όλοι ότι είναι παροχημένη αυτή η νομοθεσία πλέον από το 90. Χρειάζεται καινούργια ρύθμιση. Επίσης θεωρώ ότι είναι καλύτερο να πρόκειται για κανονισμό και όχι για οδηγία και χαίρομαι για την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή, διότι η εφαρμογή της οδηγίας η οδηγία 90 167 αυτή η οδηγία έχει σημαντικά κενά κατά την άποψή μου και δεν υπήρξε ομοιογένης εφαρμογή της ε, στα κράτη-μέλη και αυτό και προέκυψαν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η σχέση οδηγία στα διάφορα κράτη-μέλη. Και τώρα σε κάθε κράτος μέλος μπορούμε να πούμε πλέον ότι έχουμε τελείως διαφορετική προσαρμογή. Αποκλείσει σημαντικές. Επειδή είναι πολύ λεπτό το θέμα όμως, πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι πιο ομοιογενής η δράση. Άρα ο κανονισμός είναι ένα πιο αποτελεσματικό εργαλείο που θα πρέπει να εφαρμοστεί από όλα τα κράτη-μέλη με τον ίδιο τρόπο. Τώρα το να υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία για τις φαρμακοχές οτροφές και το αναφέρω και στην έκθεσή μου δεν θα πρέπει κατά την άποψή μου να οδηγήσει σε καμία διάκριση αυτή τη εναλλεκτική θεραπευτική αντιμετώπιση, δηλαδή των φαρμακούχων ζωοτροφών, έναντι οποιασδήποτε άλλη μορφή από του στόματο χορήγηση κτηνατικών φαρμάκων. Οι ζωοτροφέ θα ρυθμίζονται με το δικό τους κανονισμό, όχι άλλου είδους στόματο χορήγηση. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να συνεπάγεται διάκριση αν δεν υπάρχουν τεχνικά επιχειρήματα στα οποία να βασίζεται ή αναλυτικά επιχειρήματα που να είναι επαρκή για μια τέτοια διάκριση. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η απαιτητική σε ό,τι αφορά τη χρήση του κτηνιατρικού φαρμάκου σε όλες τις εναλλακτικές θεραπευτικές αντιμετωπίσεις. Όχι δηλαδή σε κάποιες περισσότερο από σε κάποιες άλλες ε, θεραπείες. Πάντως, και θέλω να το πω στην Κομισιόν, ότι εδώ σε αυτό το σημείο, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία μας υπέβαλε, επισημαίνω ότι υπάρχουν διακρίσεις αρνητικές σε βάρος των φαρμακούχων ζωοτροφών και υπέρ εναλλακτικών θεραπείων. Εγώ όμως πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αυστηροί. Το ίδιο για όλους τους τρόπους χορήγησης φαρμάκων, για όλες τις θεραπείες, για όλες τις εναλλακτικές η χορήγηση ενός κτηνιατρικού φαρμάκου πρέπει να διέπεται από απαιτήσει για όλες τις διαδικασίες. Στην πρόταση της Επιτροπής νομίζω ότι οι διατάξει είναι πιο αυστηρές για τις φαρμακούχες σε σχέση με άλλου είδους αποστάματος χορήγηση φαρμάκου. Τώρα, ολοκληρώνω. Σε ό,τι αφορά του ορισμούς και επειδή θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια το θέμα, θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να ορίσουμε τι τη μικροβιακή ουσία και τι εστίαται βιωτική ουσία στην νομοθεσία μας. Και πρέπει οι ορισμοί αυτοί, κατά την άποψή μου, να ενταχθούν στον πρώτο κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Οι ορισμοί δηλαδή αυτοί πρέπει να ενταχθούν στον κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Όπως συνέστησε και η κυρία Πόλσαν στη, στο σχέδιο γνωμοδότησής της. Νομίζω ότι εκεί είναι η θέση αυτών των ορισμών. Το είπε και η κυρία Πάλσεν, το εξήγησε και πολύ καλά. Αυτή είναι και η δική μου θέση και την υποστηρίζω σε αυτό το σχέδιο έκθεσης ότι στο βασικό κανονισμό πρέπει να συμπεριληφθούν αυτοί οι ορισμοί. Επίσης, Είναι σημαντικό το ζήτημα της δημόσιας υγείας, πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ παρόντες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ανησυχεί για τα ζητήματα της ε, δημόσιας υγείας, άρα η αντοχή στα, στα αντιμικροβιακές ουσίες είναι ένα ζήτημα που μας ανησυχεί. Και σχετίζεται κυρίως αυτό το πρόβλημα με την υπερβολική χρήση αντιβιωτικών για την καταπολέμηση μολύνσεων. Επομένως, αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και σε αυτόν τον οργανισμό και στους άλλους δύο που προανέφερα. Επίσης, επαναλαμβάνω ότι πρέπει αυτοί οι δύο κανονισμοί να μπουν στο βασικό κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Στην έκθεση μου όμως διευκρινίζω περισσότερο και κάποιους άλλους ορισμούς για το τι θα πει χειριστής μετακινούμενου συστήματος ανάπτυξης και τι θα πει ανάμειξη και τι θα πει συστήματος στην εκμετάλλευση. Και διευκρινίζω τον ορισμό της μη στοχευμένη ζωοτροφής, που δεν είναι πολύ σαφής. Ολοκληρώνοντας να πω ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει τις ποσότητες επιτρεπόμενες ποσότητες φαρμακών ζωοτροφών που χορηγούνται από τους παγκόσμιους κτηνοτρόφους. Ο καθορισμός χρονικών ορίων σε ένα τέτοιο κανονισμό δεν θεωρούμε ότι είναι κατάλληλος και πιστεύουμε ότι θα πρέπει ο αρμόδιος για τη συνταγογράφηση να είναι αυτός ο οποίος θα καθορίσει την ποσότητα της φαρμακούχας ζωοτροφής και το χρονικό διάστημα που απαιτείται να χορηγείται για τη θεραπεία. Γιατί ο αρμόδιος για τη συνταγογράφηση είναι ο ειδικό, ο οποίος γνωρίζει τα σχετικά με τη θεραπεία και ποιο είναι το κατάλληλότερο φάρμακο ή ποσότητα που πρέπει να χορηγηθεί. Θέλω επίση να σας πω ότι αυτό το γενικό 3% είναι επαρκές για τις δραστικές ουσίες, για όλες τις δραστικές ουσίες, τόσο αν υπάρχουν συγκεκριμένα όρια που τα οποία θα καθοριστούν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων, τα οποία θα πρέπει, αυτά δηλαδή τα όρια, τα συγκεκριμένα, τα κατώτερα δυνατά κατά την άποψή μου, θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία. Ακριβώς όπως αυτά που προβλέπονται στο κείμενο της πρότασης. Λοιπόν, έχετε πλέον την έκθεση σε, όλα, σε όλες τις γλώσσες. Είμαι στη διάθεσή σας, σας εξέχασα τα βασικότερα σημεία του κειμένου και περιμένω να ακούσω οτιδήποτε θέλετε να μου δώσετε είτε ως πληροφορία είτε ως άποψη. Ποια είναι η δική σας άποψη για την έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μπουντά είναι ο πρώτος που έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς να συγχαρώ την εισηγήτρια γιατί πραγματικά εργαστήκαμε πολύ επικοδομητικά μαζί της ως κοιόδης εισηγητές και να ευχαριστήσω επίσης και όλους όσοι συμμετείχαν στην όλη συζήτηση καθώς επίσης και σε αυτούς που διοργάνωσαν τη δημόσια κρόση που είχαμε για αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι η πρόταση αυτή θα είναι πολύ χρήσιμη και για την υγεία των ζώων αλλά σε τελευταία ανάλυση συμβάλλει και στη γενικότερη δημόσια υγεία. Υπάρχουν κάποια κρεμή ζητήματα τα οποία θα πρέπει να καλύψουμε. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε φαρμακούχες ζωοτροφές και όπως είπε και η συγγήτρια, η έκθεση αυτή συνάδει με την άλλη έκθεση που έχουμε για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Οι δύο αυτές εκθέσεις αλλοσυμπληρώνονται. Όσον αφορά όμως τις φαρμακούχες ζωοτροφές, υπάρχουν κάποιες πτυχές του ζητήματος που θα πρέπει να τις προσέξουμε όλους ιδιαιτέρως. Πρώτον, μία λογική χρήση των φαρμάκων αυτών, των ζωοτροφών αυτών. Μιλάμε για ζωοτροφές που περιέχουν ενεργά φαρμακευτικά στοιχεία. Οποιαδήποτε λοιπόν μη λογική χρησιμοποίηση των φαρμάκων αυτών μπορεί να έχει πολύ αρνητικέ επιπτώσει. Δεν αναφέρομαι βέβαια μόνο στα αντιβιωτικά. Τα αντιβιωτικά δεν είναι τα μόνα τα οποία δημιουργούν αντοχή. Πολλά φάρμακα μετά από μακροχρόνια χορήγηση μπορούν να δημιουργήσουν υψηλά επίπεδα αντοχή τόσο στον, στο ζώο και συνέχεια αυτό να περάσει και στον άνθρωπο. Πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι φαρμακούχε αυτέ οτροφέ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προληπτικά γιατί αυτό μπορεί να έχει, όπως σας είπε επιζήμιες επιπτώσεις στην υγεία των ζώων και των ανθρώπων και θα πρέπει να είναι σαφές πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά, όλες αυτές τις φαρμακούχες ζωοτροφές για το σύνολο και τις ομάδες ζώων. Και να φέρουμε εδώ πέρα στα χειροειδή, στα πουλερικά, θα πρέπει να χορηγούμε τη θεραπεία αυτή σε ομάδες ζώων μόνο όταν πραγματικά το έχουν ανάγκη τα ζώα. Ξέρουμε ότι μερικές φορές ορισμένα ζώα μπορούν να παρουσιάζουν κάποια κλινικά ή προκλινικά συμπτώματα και είναι ο γιατρός ο υπεύθυνο ο οποίος θα πρέπει να αποφασίσει ποια φάρμακα θα δοθούν και για ποιο χρονικό διάστημα. Επίσης, να αναφερθούμε και στις ζωογειονομικές συνθήκες Ξέρετε ότι υπάρχουν ορισμένοι που θα ήθελαν να χρησιμοποιούν τις φαρμακούχες ζωοτροφές προκειμένου να αντισταθμίσουν κάποια κενά τα οποία μπορούν να υπάρχουν στην όλη διαχείριση της υγείας των ζώων στα πλαίσια ενός αγροκτήματος. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε μια τόσο υπερβολική χρήση. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα πραγματικό δικό χάρτη, χρειαζόμαστε πραγματική χνηλασιμότητα των φαρμακούχων ζωοτροφών, Αρμόδιος θα πρέπει να είναι ο αρμόδιος συνταχογράφησης και θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται και στην αγροτική εκμετάλλευση αλλά και τι γίνεται με τα φάρμακα αυτά όταν τελικά δεν χρησιμοποιούνται, όταν τελικά δεν χορηγούνται στα ζώα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα νομικό μέσο το οποίο θα είναι πραγματικά χρήσιμο για όλους εμπλεκομένους. Οι σκιοαντισηγητές ε, θα έχουν 2,5 λεπτά και όλοι οι άλλοι ομιλητές 1,5 λεπτό. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Και το λόγο έχει η κυρία Γκέρινγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να πω ευχαριστώ στον εισηγητή, ε, στην εισηγητρία. Ήταν πολύ μεγάλη ευχαρίστηση η κουβέντα μαζί τη, ε, πολύ ανοιχτή, πολύ ειλικρινή. Ε, χαιρετίζω λοιπόν την έκθεση γιατί είναι ένα θαυμάσιο σημείο εκκίνηση ε, και θέλω να πω ότι συμφωνώ με τις και εγώ ανησυχώ όσον αφορά το σαφή διαχωρισμό, όσον αφορά του στόχους αυτού του κανονισμού και του κανονισμού για τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Ε, πράγματι ε, θα πρέπει να υπάρχουν ε, κάποιες, κάποιοι ορισμοί, να διευκρινιστούν ορισμοί, αλλά υπάρχουν και θέματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε. κυρίως όσον αφορά τα ιατρικά φάρμακα. Ε, θεωρώ ότι θα πρέπει την έκθεση αυτή και τις δύο να τις διατηρήσουμε γιατί αντιμετωπίζουν διαφορετικά θέματα. Και νομίζω πρέπει να είναι σαφές ότι εδώ μιλάμε για φαρμακούχες ζωοτροφές, μιλάμε και για στοιχεία που έχουν άμεση σχέση με τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Χαίρομαι που έγινε η δεκτή πρότασή μας ε, να αφαιρεθεί αυτό το κομμάτι που είχαμε προτείνει γιατί δεν θα ωφελούσε κανέναν. Παραμένουμε λοιπόν στο 3% ε, το οποίο είναι πιο κατάλληλο και αν αυτό αλλάξει νομίζω ότι θα πρέπει να κατατεθούν και συγκεκριμένες προτάσεις που να έχουν εγκριθεί από την ΕΦΣΑ. Να γνωρίζουμε δηλαδή όλοι λειτουργούμε με βάση επιστημονικές μελέτες και όχι τυχαία, τυχαίους αριθμούς. Η πρόταση Κομισιόν καθορίζει την, ε, το όριο για, σχετικά με τις συνταγογραφήσεις Υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που θέλουν να υπάρχουν στην τελική έκθεση. Αυτά τα έχω καλύψει στις τροπολογίες μου και τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι να διασφαλίσουμε ότι οι αρμόδιοι STPs λέγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν είναι κτηνίατροι ε, να μπορούν αυτοί να συνταγογραφούν σε βαθμό βέβαια που κάτι τέτοιο γίνεται αποδεκτό από την εθνική νομοθεσία. Αυτό συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, εάν περιοριστεί αυτή η δυνατότητα αυτό θα είναι εις βάρους της υγείας των ζώων. Ε, θεωρώ ότι βέβαια αυτό δεν είναι τόσο επίγον το θέμα για την εισηγήτρια, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε την καλοσύνη να δεχτεί ότι αυτό είναι πρόβλημα γιατί το δικό μου το κράτος, τη δική μου τη χώρα και ξέρω ότι μπορώ να υπολογίζω στην υποστήριξή της. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φέντερλι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τη συζήτηση και ακούσαμε ότι πολλοί κατανόησαν το πόσο σημαντικό είναι το να μην υπάρχει ε, υπερβολική χορήγηση φαρμάκων στα ζώα, γιατί αυτό μπορεί να βλάψει και τα ζώα. Επίσης ε, στην Επιτροπή μας βιώσαμε ότι μπορεί να υπάρξει αντίδραση στα βακτήρια ε, και να φυγούν τα ζώα. Υπάρχουν ζώα τα οποία ε, δεν θα γίνουν καλύτερα, δεν θα γίνουν καλά, δεν θα αποκτήσουν την υγεία τους από τη χορήγηση αντιβιωτικών. Βλέπουμε, έχουμε ακούσει με αριθμούς, 25.000 άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο ε, πεθαίνουν από αυτή την αντίδραση στα ε, αντιβιωτικά. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι δυσάρεστο γεγονός ότι η συγγήτρια δεν μιλάει περισσότερο για την προληπτική χρήση Βεβαίως ε, πρέπει να εξετάζουμε και διάφορες, ε, διάφορα είδη ζώων, αλλά ε, υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί μία ασθένεια. Βεβαίως τα αντιβιωτικά χρησιμοποιούνται πολλές φορές προληπτικά παρά ειδικά για μια ασθένεια και υπάρχει ένα είδος αντιβιωτικής ομπρέλας θα λέγαμε που σημαίνει ότι δεν είναι αρκετά καλή η κτηνοτροφία. Όσον αφορά ε, το πρώτο θέμα σχετικά με την υγεία των, υγεία ζώων, νομίζω ότι αυτό το σημείο καθορίζει τη βάση για το πώς πρέπει να σκεφτούμε στο μέλλον. Ε, και κατόπιν θα δούμε ε, πώς θα εξετάσει το θέμα των ε, φαρμακούχων ζωοτροφών. Πιστεύω ότι η Κομισιόν στο μέλλον πρέπει να κάνει περισσότερα πράγματα. Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο μετά από αυτή την πολιτική που τελειώνει αυτό του, αυτού του έτους. Να ασκήσουμε πίεση γιατί αλλιώς δεν θα εκπονηθεί η απαραίτητη νομοθεσία. Εξάλλου, αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η ομαδική θεραπεία. Ε, υπάρχει μόνο περιορισμός ε, στη συνταγογράφηση. Εγώ όμως θεωρώ ότι αυτό είναι ο μόνος δρόμος ο σωστός αν θέλουμε να υπάρχει πραγματική αντίδραση στα ε, αντιβιωτικά. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που τελικά καταφέρνουμε να έχουμε αυτή τη συζήτηση σε ολόκληρη την Ευρώπη για τους κινδύνους που σχετίζονται με την υπερβολική χρήση αντιβιωτικών. Ο τομέας του φαρμάκου στην Ευρώπη συνολικά αλλά και η ιατρική κοινότητα επισημαίνει τους κινδύνους και για την ανθρώπινη υγεία αλλά και για την υγεία των ζώων. Ήδη σήμερα έχουμε χιλιάδες άτομα που όπως το βλέπουμε στα νοσοκομεία ή αλλού, υποφέρουν από το ζήτημα αυτό της μικροβιακής αντοχής. Και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πρόταση. Η κυρία Πάλσεν έχει εργαστεί πολύ καλά για το φάκελο αυτό. Και σίγουρα μπορούμε να δράσουμε και εμείς για να περιορίσουμε ώστε να τον περισσότερο αυτό το πρόβλημα. Έχοντας υπόψη λοιπόν τη σημερινή κατάσταση, Πρέπει να πω ότι λυπάμαι. Που βλέπουμε εδώ σε αυτό το σχέδιο έκθεσης μια προσπάθεια μείωσης κάποιων ορίων ε, της ε, Κομισιόν. Βλέπω να εισάγονται κάποιες εξαιρέσεις. Είναι επιβάλλονται λιγότερο αυστηριόροι για τη χρήση φαρμάκων και ποιο είναι ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στη χωρίς δύο δόσεων του φαρμάκου και του καθεξής. Με αντιβιωτικά. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να προβούμε σε προληπτικές ενέργειες για να γνωρίζουμε αν έχει κίνδυνο η χρήση των αντιβιωτικών ή από τη στιγμή που ακολουθούνται ε, κακές πρακτικές, τι θα πρέπει να γίνει. Είναι ένα ηθικό σκάνδαλο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακολουθήσουμε αυτήν την οδό όταν παντού σχεδόν γίνεται ε, δημόσια συζήτηση και ο πληθυσμό ανησυχεί, ο κόσμος ανησυχεί για την γενικευμένη χρήση αντιβιωτικών. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μας απασχολήσει το ζήτημα επαρκώς και θα αποφύγουμε να αποδυναμώσουμε όλες τις προτάσεις Κομισιόν. Um, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. με τον κίνδυνο να επαναλάβω αυτά που είπαν ε, οι υπόλοιποι, θεωρώ ότι το σημαντικότερο σημείο της συζήτησης που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι το ότι έχουμε καταφέρει να αποκομίσουμε πάρα πολλά διδάγματα για το πώς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το μέσο αυτό το νομοθετικό για να εξορροπήσουμε κάπως τα πράγματα. Προστασία δηλαδή των ζώων αφενός και εμπορική διάθεση όλων αυτών των ουσιών αφετέρου. Κυρίως όμως νομίζω ότι η βασική μας προτεραιότητα πρέπει να είναι η ανθρώπινη υγεία, η υγεία των ανθρώπων. Και πιστεύω ότι εδώ πέρα υπάρχει ακόμα ένα περιθώριο βελτίωσης σε αυτό το σχέδιο έκθεσης. Διότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η αρχή ε, της πρόληψης θα περιλαμβάνεται στην διαδικασία που θα ακολουθήσουμε. Γιατί ξέρουμε ότι η αντοχή στα αντιβιωτικά και η μικροβιακή αντοχή είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάζει αύξηση παντού στην Ευρώπη και αυξάνεται όλο και περισσότερο και πολύ πιο γρήγορα σε όλες εκείνες τις περιοχές της Ευρώπης όπου δεν υπάρχουν απαραίτητες ρυθμίσεις. Από την άλλη βέβαια καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε στο σημείο εκείνο που οι κτηνοτρόφοι, οι γεωργοί θα είναι σε θέση να δίνουν εξατομικευμένα, αν θέλετε, εντελώ ξεχωριστά σε κάθε ζώο ξεχωριστά το φάρμακο το οποίο πρέπει να χορηγηθεί στο ζώο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι ιδίω για κάποιε μικρέ εκμεταλλεύσει που δεν έχουν του απαραίτητου πόρου είναι πολύ δύσκολο να γίνει μια τέτοια εξατομικευμένη θεραπεία. Τούτων λεχθέντων Ξέρω ότι ε, αν δεν καταφέρουμε και στα πλαίσια της συμφωνίας TTIP να διευθετήσουμε τα ζητήματα αυτά, δεν θα πάμε πάρα πολύ μακριά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αν θέσουμε τα απαραίτητα χέγγια για τις φαρμακούχες ζωοτροφές στην Ευρώπη, δεν κάνουμε σπουδαία πράγματα αν για το χοιρινό, το βοδινό ή άλλους τύπους κρέατος από τις ΗΠΑ δεν ισχύουν οι ίδιες διασφαλίσεις, δεν ισχύουν τα ίδια κριτήρια. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν ε, τελείωσε η συζήτηση για αυτό το θέμα. Και όλοι οι επόμενοι ε, ομιλητέ θα έχουν δυνατόν να μιλήσουν για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Κυρία Γιούσο, πράγματι όπως είπε και η συγγύτρια, είναι πολύ σημαντικός αυτός ο κανονισμός και θα ήθελα να συγχαρώ πρώτα απ' όλα την συγγύτρια, διότι Κάνει εξαιρετική δουλειά και βελτίωσε σημαντικά την πρόταση της Κομισιόν σε πολλές πτυχές. Θα αναφερθώ σε ορισμένες εξ αυτών. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός ο καθορισμός ε, μέγιστον ορίων ε, διασταυρούμενης επιμόλυνσης, όπως τα λέμε, των δραστικών ουσιών, γιατί η Κομισιόν εδώ μας προτείνει 1%. Δεν υπάρχει καμία όμως επιστημονική βάση για το 1 Άρα η ΕΦΣΑ πράγματι θα πρέπει να είναι η αρχή που θα ορίσει αν αυτό είναι σκόπιμο, εφικτό και ποιο ποσοστό θα πρέπει να καθοριστεί. Το 3% νομίζω για τις δραστικές που προτείνει η συγκήτρια ως ποσοστό μεταφοράς είναι ένα καλό ποσοστό. Σε ό,τι αφορά τώρα την αποθήκευση ή την εκ των προτέρων παραγωγή. Η Κομισιόν απαγορεύει και τα δύο, και την εκ των προτέρων παραγωγή και την αποθήκευση φαρμακούχων ζωοτροφών. Αυτό όμως θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ε, των ομάδων ζώων ίσων ε, σημασίας, ε, όπως λέγονται. Δεν έχω το χρόνο να σας εξηγήσω ε, τις λεπτομέρειες, αλλά εν γέννη πρέπει να πω ότι η έκθεση είναι πολύ καλή. Ευχαριστώ. Η συγγήτρια μας είπε ότι θα ήθελε πάρα πολύ να δει ένα κανονισμό. Εγώ δεν είμαι καθόλου ενθουσιώδης για το να έχουμε κανονισμό στον τομέα αυτό. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί κανονισμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή όσον αφορά το ζήτημα αυτό των φαρμακούχων ζωοτροφών. Οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η παραγωγή ζωοτροφών βάζουν αυτό το φάρμακο στις ζωοτροφές και αυτό είναι ουσιαστικά μια χάρη που κάνουν στους πελάτες τους. Καταλαβαίνετε ότι η ίδια διαργασία αυτή είναι πάρα πολύ επαχθής για αυτούς. Αν υπάρχουν επιπλέον και περισσότεροι κανόνες, καταλαβαίνετε ότι θα εγκαταλείψουν εντελώς την, το, το όλο εγχείρημα. Επομένως θα βάλει κατά του όλου κλάδου. Αν δούμε το άρθρο 5 παράγραφος 2 δέλτα, μιλάμε για το ψευδάργυρο. Ο ψευδάργυρος είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να προσθεθεί στα τρόφιμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όμως και ως φάρμακο. Εμείς το επιλύσαμε στη Βρετανική νομοθεσία αυτό το πρόβλημα, επομένως το άρθρο 5 στον προτινόμενο κανονισμό ενδεχομένως να μας γυρίσει πίσω και να μπερδέψει τα πράγματα. Επίσης το άρθρο 7 όσον αφορά την μεταφορά. Ξέρετε ότι η Στομοσπονδία των Γεωργικών Βιομηχανιών δεν χρησιμοποιεί μια πολύ ισχυρή διατύπωση συνήθω, αλλά εν προκειμένου έχει πει ότι είναι παράλογη η πρόταση αυτή, δηλαδή δεν πρόκειται στην πράξη να λειτουργήσει. Σα παρακαλώ λοιπόν πολύ, σα το λέω ότι εγώ έχοντα εμπειρία αγρότη δεν πρόκειται η πρόταση αυτή να λειτουργήσει στην πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ε, θέλω να ευχαριστήσω γιατί μέχρι τώρα συνεργασία με την συγγήτρια. Επίσης ε, να ευχαριστώ πολύ για το σχέδιο της έκθεσης και θέλω να ευχαριστήσω για το ότι προσαρμόσαμε ε, το χρονοδιάγραμμα ανάμεσα στον κανονισμό για τα φάρμακα και τον κανονισμό για, τα, φαρμακού, για τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Νομίζω ότι το στόχο μας τον επιτύχουμε με τον καλύτερο τρόπο αν τελικά πράγματι συνδυάσουμε αυτές τις δύο εκθέσεις. Θέλω να πω όμως ότι υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες όπου πιστεύω ότι δίστανται οι απόψεις. Χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι καταλήξαμε τους ορισμούς σε συνδυασμό με την κυρία Γκροστέτ ε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ορισμός ε, της προφύλαξης, ε, της θεραπευτικής χρήσης των μειγμάτων. Νομίζω ότι αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ σημαντικά. Και κατά τα άλλο θέλω να επισημάνω ότι όσον αφορά τον κίνδυνο μετακύλησης, υπάρχει αυτό το 3% αλλά δεν βασίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά όσον αφορά στα αντιβιωτικά και σε άλλες δραστικές ουσίες. Θα ψηφίσουμε αύριο και θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν στη συζήτηση που θα ακολουθούσε θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη και οι δικές μου παρατηρήσεις. Ο κύριος Δαντά, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το κείμενο αυτό να καθορίσει ξεκάθαρα κάποιες θεματικές ενότητες που έχουν να κάνουν και με την ομολογία που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το... Η έκθεση αυτή σχετίζεται άμεσα με την έκθεση για τα κτηνιατρικά φάρμακα, αλλά σχετίζεται επίσης και με το ζήτημα της δημόσιας υγείας, συνεπώς η συγγήτριά μας εδώ πέρα νομίζω ότι κρατάει μια απόσταση σε σχέση με τις θέσεις του Συμβουλίου και νομίζω ότι υπερβαίνει εδώ πέρα κάποια όρια. Εμείς ε, νομίζω ότι θα πρέπει να συνταχθούμε λίγο με αυτό που μας ζητάνε οι ίδιοι επαγγελματίες του τομέα. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί προκειμένου να μην υπάρχει καμία περαιτέρω διάδοση των αρνητικών επιπτώσεων μιας υπερβολικής χρήσης τέτοιων φαρμακούχων ζωοτροφών. Θα ήθελα λοιπόν σχετικά με τα ζητήματα αυτά να καταθέσω και μια σειρά από τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να πω ότι την έκθεση την βρίσκω πολύ ρεαλιστική, σωστά τη σκέφτηκε η συντάκτρια και σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή. Έχω όμως ε, κάποιες ερωτήσεις, έστω και αν ε, συζητήσαμε διεξοδικά τα διάφορα θέματα. Δηλαδή, ε, πρέπει να είναι πιο σαφείς οι ορισμοί που υπάρχουν στην οδηγία. Για τη τελική ανάλυση πρόκειται για την έκθεση της κυρίας Πάουσεν. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε σύγχυση για το, την περιεκτικότητα των ουσιών που περιλαμβάνονται στις φαρμακούχες τροφές. Το σελιντόν, παραδείγματος χάνει, θεωρείται αντιβιωτικό, όμως προέρχεται από την κατηγορία των ε, φυτικών φαρμάκων, προέρχεται από φυτά δηλαδή. 0,01% είναι το όριο για να μπορεί να γίνει ο έλεγχος και αυτό σημαίνει ότι τιμωρούνται οι παραγωγοί ζωοτροφών οποτεδήποτε υπάρχει η εντοπιστή αυτή η ουσία στις ζωοτροφές. Σε άλλες όμως χώρες το ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο. Άρα δηλαδή θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς ποιοι είναι οι ορισμοί που ισχύουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Ε, και ευχαριστώ την εισηγητριά μας. Επιτρέψτε μου κάποιες παρατηρήσεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν εγκρίσεις και για λιγότερο από ε, τα δύο γραμμάρια ανατόνο. Κυρίως ε, όσον αφορά την ε, προσαρμογή στο μέγεθος των ζώων. Γιατί στα κράτη-μέλη έχουμε και μικρές ε, και μεγάλες ε, κτηνιατρικές μονάδες. Και θέλω να επισημάνω ότι οι μίκτες, οι κινητοί μίκτες όπως είναι γνωστοί σε ορισμένα κράτη-μέλη, αυτή είναι πολύ σημαντική. Σε μένα, παραδείγματο παραδείγματος υπάρχουν μικρές ε, δομές ε, ή αν θέλετε οι γεωργοί ε, παράγουν επιτόπου τις τροφές και δεν τις αγοράζουν. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να ε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα να μπορούν να πηγαίνουν σε ένα μίκτη και να υπάρχουν και κινητές μηχανές μίξης θα ήθελα λοιπόν ε, να το λάβετε αυτό ε, στις ε, συζητήσεις που θα ακολουθήσουν. Κύριε Μαγκίνες, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Και επειδή έχει μια ακρόαση για την αλυσίδα προμήθειας τροφίμων, άργησα να έρθω. Στο συγγνώμη, τρία σημεία θέλω να αναφέρω. Ορισμένα εξ αυτών αναφέρθηκαν όπως το 1% η συγγήτρια την οποία θέλω να ευχαριστήσω, νομίζω το έλυσα το ζήτημα. Η συζήτηση τώρα για τους αρμόδιους, εκτινο, κτηνίατος και και αυτό καλύφθηκε από τους προλαλήσαντες. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στο κείμενο. Θα καταθέσω τροπολογίες, παραδείγματος χάρη για τη χρήση συγκεκριμένων ουσιών ή ε, δραστικών ουσιών. Πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τους όρους ε, και επίσης ένα θέμα είναι το διασυνοριακό εμπόριο φαρμακούχων ζωοτροφών ε, και γι' αυτό θα καταθέσω τροπολογίες. Θέλω πάντως να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Το θέμα είναι σημαντικό, ίσως πιο σημαντικό σε κάποια άλλα κράτη μέλη από ό,τι σε άλλα έχουν άλλωστε διαφορετική μεταχείριση τα κράτη-μέλη των άρρωστων ζώων. Σε άλλα χρησιμοποιούνται πολύ πιο πολύ οι φαρμακούχες ζωοτροφές, σε άλλα λιγότερα. Τα άρθρα που με ενδιαφέρουν περισσότερο πάντως και τα οποία θα καταθέσω τροπολογίες είναι τα άρθρα 11, 7 και 5, 2. Hm. Äh, και εγώ ευχαριστώ θερμά την εισηγήτρια. Ε, να κάνω δύο ερωτήσεις. Εδώ πρόκειται για την κρίση φαρμακούχων ζωοτροφών και η κοινή γνώμη ενδιαφέρεται ιδιαίτερα. Κυρίως όσον αφορά και την ε, χρήση αντιβιωτικών. Και ρωτώ, καταστήσαμε σαφές ότι εδώ είμαστε υπέρ της στρατηγικής ελαχιστοποίησης. Δηλαδή, όσο λιγότερα αντιβιωτικά, τόσο καλύτερα. Και κάτι άλλο. Στα αντιβιωτικά ε, δεν θα πρέπει να παραιτηθούμε από 7 ως προς τη χρήση του στις ζωοτροφές ή μήπως ε, υπάρχουν ε, αντιβιωτικά ε, που, είναι, που δεν επιτρέπουν τη διείσδυση νερού. Εγώ ξέρω ότι όλα τα αντιβιωτικά επιτρέπουν την διείσδυση νερού. Όλα αυτά στην δική μου την περιοχή όπου ζω αυτή τη στιγμή είναι στην, ε, στους πηχαίους των και παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω και εγώ ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους ορισμούς στο κείμενο αυτό, όπως ο κύριος Λίνς και οι υπόλοιποι σκιώδεις ηγητές, έτσι και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε πρώτα ποια θα είναι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Στη γνωμοδότηση αυτή νομίζω θα πρέπει να επικεντρωθούμε στους ορισμούς. Ο κύριος Γιάρα αναφέρθηκε επίσης στα αντιβιωτικά και στη χρήση τους. Να επιμείνω και στο ζήτημα αυτό. Ξέρετε ότι ο ΩΣΑ μας έχει πει ότι πολύ σύντομα θα έχουμε μία αύξηση της τάξης του 67% όσον αφορά τη χρήση των αντιβιωτικών παντού στον κόσμο. Και από ό,τι φαίνεται θα αυξηθεί παράλληλα και η κατανάλωση κρέατος, που ενδεχομένω να εμπεριέχει τέτοια αντιβιωτικά. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να προβλέψουμε μια δραστική μείωση των αντιβιωτικών και μια καλύτερη διαχείριση των αντιβιωτικών από τις επιχειρήσεις τις γεωργικές. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τιμωρούμε τους αγρότες, τους παραγωγούς επειδή δεν είναι πλέον ανταγωνιστικοί. Νομίζω ότι θα πρέπει από κοινού παγκοσμίω να γίνει μια προσπάθεια για τη μείωση της χρήσης αντιβιωτικών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντέση έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια και θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που μόλις τώρα ελέγχθη. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει υγιής διατροφή των ζώων και γι' αυτό είναι απαραίτητα τα φάρμακα. Αλλά ε, όπως και οι άνθρωποι και τα ζώα αρρωσταίνουν και εκεί κάτι πρέπει να γίνει. Στη Γερμανία λοιπόν κάναμε έναν έλεγχο. Ε, ήρθε και με βρήκε ο πρόεδρος των Ευρωπαίων ε, κτηνιάτρων Γάλλος και μου είπε θέλει το σύστημα να επεκταθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε τη δυνατότητα δεκμηρίωση, τη δυνατότητα ίχνη λασιμότητας. Να δούμε πού έχουν χρησιμοποιηθεί πια αντιβιωτικά. Και έτσι μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλο και λιγότερα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχουμε το στόχο μας, να ακολουθήσουμε τη σωστή κατεύθυνση. Πρόεδρος, και τώρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Πομελίνη. Bardzo proszę przedstawiciela komisji, panią Pongelini. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν, παρακαλώ πολύ. Πρώτα απ' όλα κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την συντάκτρια για τη δουλειά της, γιατί πρέπει να σας πω ότι πράγματι ε, αυτά όλα τα θέματα που συζητάμε είναι πολύ τεχνικά και πολύ δύσκολα. Λοιπόν, όσον αφορά την πρόταση που λάβαμε και μετά από τη συζήτηση που είχαμε μέχρι τώρα, μετά από τα δύο αυτά, θέλω να πω ότι οι προτάσεις που έχουν ε, γίνει είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ σημαντικές. Όλοι νομίζω συμφωνούμε επί του γεγονότος ότι ο κοινός στόχος του κανονισμού της πρότασης είναι να προστατευτεί η υγεία των ζώων μας και βεβαίως παράλληλα να προστατευτεί και η υγεία των ανθρώπων με στόχο να αντιμετωπίσουμε αυτό το νέο κίνδυνο που μοιάζει να παραμονεύει ε, που είναι η αντίδραση, η αντοχή στα ε, ε, αντιβιωτικά. Αυτή λοιπόν είναι η γραμμή που ακολουθούμε και η δική μας η πρόταση είναι να επιτύχουμε, να επιδιώξουμε την ισορροπία ανάμεσα αφενός στην χρήση αντιβιωτικών για να προστατεύσουμε την υγεία των ζώων και αφετέρου στην αναγκαιότητα να μειώνεται η χρήση των αντιβιωτικών ακριβώς για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ε, αντοχής στα αντιβιωτικά, κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο τα ζώα, αφορά και τους ανθρώπους. Ε, οι οποίοι και αυτοί αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Άκουσα λοιπόν ότι ορισμένοι ευρωβουλευτές έχουν δυσκολία στο να δεχτούν κάποιους περιορισμούς, όμως ας μην ξεχνάμε ότι ο στόχος είναι ακριβώς αυτός, να επιτύχουμε ισορροπία. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος, ισορροπία για να μπορούμε με τον τρόπο αυτό να προστατεύσουμε γενικότερα την δημόσια υγεία. Για να επιτύχουμε λοιπόν το στόχο μας, επιβάλαμε ε, όρια στην cross-contamination. Ε, γνωρίζουμε ότι αυτό είναι βέβαια κάτι που θα πρέπει να το επανεξετάσουμε, να δούμε λιγάκι τα όρια που έχουμε καθορίσει κάτω από το πρίσμα των προτάσεων αλλά και άλλων συζητήσεων που έχουν γίνει στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να έχουμε βέβαια κατά νου ότι δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τη φιλοδοξία μας που είναι να αποφύγουμε αυτή την ε, ε, μόλυνση, την cross-contamination. Άρα δηλαδή η ενδιάμεση λύση είναι ακριβώς να ορίσουμε κάποια όρια για να αποφύγουμε όπως σας είπα την διασταυρούμενη επιμόλυνση, την cross-contamination. Και αυτό που μας ενδιαφέρει επίσης είναι να ε, εντοπίσουμε ε, και συγκεκριμένες προτάσεις που θα βασίζονται στα στοιχεία της ΕΦΣΑ. Αυτή λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος μας. Κατόπιν υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που έχουν ε, σχέση με τους ορισμούς, θέματα τα οποία έχουν θίξει οι βουλευτές, δηλαδή κάποιες διευκρινήσεις για το πώς ακριβώς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ορισμοί. Αυτό νομίζω ότι περιλαμβάνονται και στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί για την έκθεση. Στις δικές μας προτάσεις, εμείς έχουμε κάποιες ε, παρατηρήσεις να κάνουμε με την έννοια ότι η χρήση της ε, δραστικής ουσίας ή του, ε, των φαρμακευτικών ζωοτροφών, αυτό δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι διαφορετικά πράγματα. Με την έννοια ότι και οι χρήσεις είναι διαφορετικές. Εδώ λοιπόν αναφέρομαι και σε μια άλλη παρατήρηση που έγινε, η οποία είναι ότι μιλάμε τελικά για φάρμακα, μιλάμε για ζωοτροφές που περιλαμβάνουν ε, φαρμακούχες ουσίες για να επιτευχθεί ο στόχος μας. Άρα δηλαδή ο η χρήση πρέπει να γίνεται δια του στόματος και αυτό για ειδικέ περιπτώσεις ζώων. Ενώ όπως υπόθηκε και εδώ σήμερα το πρωί, ή τώρα το απόγευμα σχολή κατά τη διάρκεια δηλαδή της συζήτησης, η τωρα το απογευμα σχολη κατα τη συζητηση η θεραπεια με ζω, φαρμακούχες ζωοτροφές γίνεται δηλαδή ε, με ουσίες ε, ε, που αφορούν όμως ένα συγκεκριμένο ζώο. Γιατί όταν πρόκειται για ομάδες, εκεί μιλάμε για διαφορετική προσέγγιση. Εγώ εκείνο το οποίο θέλω να πω και με αυτό κλείνω είναι ότι κατά την άποψή μου ο στόχος είναι κοινός για όλους. Δηλαδή η προστασία της δημόσιας υγείας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να εντοπίσουμε τα μέσα για να επιτύχουμε το στόχο μας. Ε, μερικές προτάσεις που έγιναν ε, συμφωνούμε από αυτόν. Ε, σε άλλες πάλι περιπτώσεις θεωρώ ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα, να δούμε καλύτερα τι είναι τελικά εκείνο που επιδιώκουμε. Θα έλεγα λοιπόν ως πρώτη προσέγγιση, η πρώτη προσέγγιση είναι απόλυτα ικανοποιητική και νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς, αλλά σύντομα παρακαλώ, κύριε Συγητρία. Ναι, το μόνο που έχω να προσθέσω στην πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων είναι να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για τις παρεμβάσεις. Έχουμε κοινού στόχους, νομίζω όλοι. Συμφωνούμε από των στόχων, επομένως είμαι στη διάθεσή σας για να έχουμε τελικά έναν κανονισμό στον τον καλύτερο Δεν ξέρω αν το γερμανικό μοντέλο, κύριε Ντές, είναι το ότι καλύτερο. Όπως και αν έχει όμως, σίγουρα. Για να πετύχουμε τους στόχους και για να περιορίσουμε τις διαστάσεις του φαινομένου της μικροβιακής αντοχής ή της αντοχής στα αντιβιωτικά, θα πρέπει να εγκριθεί ένας κανονισμός για να εφαρμοστεί από όλα τα κράτη-μέλη Είμαι στη διάθεση όλων των συναδέλφων για να εργαστούμε από κοινού και να βελτιώσουμε την έκθεση για να φτάσουμε στον κανονισμό που είναι πολύ σημαντικός. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όπως ξέρετε, η συντάκτρια της έκθεσης μετά από διαβούλευση με τους υπόλοιπους συναντέλφους αποφάσισε να αναβληθεί ε, για το φθινόπωρο η ψηφοφορία. Μέχρι τις 21 Ιουνίου έχουμε την καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση τροπολογιών. Στην ε, Ολομέλεια ε, θα ψηφίσουμε τον Νοέμβρη. Ευχαριστούμε λοιπόν τη συντάκτρια, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και τώρα πάμε στο τέταρτο σημείο τη σημερινή διάταξη που είναι η υγεία των ζώων. Η κυρία Πάουλσεν είναι η συντάκτρια της έκθεσης και έχουμε πολύ καλά νέα. Επικράτησε συμφωνία όσον αφορά την σχετικά με την υγεία των ζώων έγιναν συζητήσεις με το Συμβούλιο. Σας συγχαίρω λοιπόν κυρία Συγήτρια και σας ευχαριστούμε θερμά για την ε, πολύ καλή σας δουλειά. Νομίζω λοιπόν ότι μπορώ ήδη τώρα να σας δώσω το λόγο θα, μα θα μας παρουσιάσετε τα αποτελέσματα του τριμερού διαλόγου και παρακαλώ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όντως την πρώτη η είχαμε τον τελικό τριμερή διάλογο για αυτόν τον νέο κανονισμό για την υγεία των ζώων ο οποίος ε, φέρει άλλο όνομα πλέον και ονομάζεται Κανονισμός για την πρόληψη και τον έλεγχο των μεταδοτικών ασθενειών και ουσιαστικά αυτή είναι η βάση, αν θέλετε, του νέου αυτού κανονισμού και επ' αυτού είχαμε και πολιτική συμφωνία. Η πολιτική συμφωνία δεν προβλέπει τίποτα παραπάνω από το να καταφέρουμε τελικά να περιορίσουμε αυτές τις μεταδοτικές ζωικές νόσους και αυτό ουσιαστικά αποτελεί πραγματικό επίτευγμα της Επιτροπής μας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν πολύ μεγάλη λοιπόν η νίκη και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και θα του ευχαριστήσω πάρα πολλές φορές βασικά για την καταπληκτική συνεργασία που είχαμε. Η κυρία Μπαγκούτς επίσης και η Ελίζα Πεθιέκλε ήταν παρούσες στο πρώτο τμήμα της όλης αυτής διαδικασίας, πριν γίνει δηλαδή πρώτη ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Τα όσα κάναμε τότε στη φάση εκείνη καθόρισαν το ότι μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα ιδιαίτερα πολύπλοκο και καταφέραμε να εστιαστούμε στους βασικούς στόχους και τις βασικές αρχές πίσω από τον κανονισμό αυτό. Αυτή τη στιγμή πετύχαμε κοινή συμφωνία για τους στόχους και τις αρχές. Τα πράγματα κύλησαν πολύ πιο ομαλά και πολύ πιο γρήγορα όταν αρχίζαμε να χτενίζουμε δηλαδή το κείμενο προκειμένου να το κάνουμε ένα συνάδει με αυτούς τους βασικούς στόχους και τις βασικές αυτές αρχές. Σας ε, συνιστώ λοιπόν και εσείς κάθε φορά που αντιμετωπίζετε πολύπλοκα ζητήματα να ξεκινάτε με αυτή τη μέθοδο εργασίας. Καθορισμός στόχος και αρχών και έπειτα εξέταση του κειμένου. Έγινε λοιπόν η πρώτη ψηφοφορία 570 υπέρ στην Ολομέλεια και στη συνέχεια δόθηκε σε μένα και στους πιο δυσηγητές μια πολύ ηγετική θέση στους τριμερείς διαλόγους που συζητήθηκαν ακριβώς επειδή είχαμε μια πολύ δυνατή εντολή που μας δόθηκε από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό δίδαγμα, να καταφέρνουμε κάθε φορά να πετυχαίνουμε συμβιβασμούς και να συσπυρωνόμαστε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε φορά που βρίσκουμε απέναντί μας το, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε ότι όταν είμαστε διαιρεμένοι είμαστε και αδύναμοι, όταν είμαστε όμως ενωμένοι είμαστε πολύ πιο ισχυροί. Το πιο σημαντικό νέο στοιχείο που προέκυψε από την νέα, από την πρώτη με συγχωρείτε ψηφοφορία είναι ότι η ευημερία των ζώων, η καλή διαβίωση των ζώων συνδέεται πλέον με την ίδια την υγεία των ζώων και με το ζήτημα της μικροβιοκής αντοχής. Είναι πολύ σημαντικό το ότι οι τρεις αυτές έννοιες πλέον συνδέθηκαν στον κανονισμό. Και βλέπουμε ότι υπάρχει και μια πιο έντονη πολιτική απήχηση πλέον για τα ζητήματα αυτά μετά την υποβολή της έκθεσης 24 Απριλίου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πάντως για πρώτη φορά έχουμε μία νομοθεσία η οποία διασυνδέει άμεσα την υγεία των ζώων, την καλή διαβίωση των ζώων και την ανθρώπινη υγεία. Η νέα λοιπόν αυτή νομοθεσία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου στην ε, καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής τόσο για τα ζώα όσο και για τους ανθρώπους. Και βέβαια θα έχει πολύ θετικέ συνέπειες και για το ίδιο το περιβάλλον. Ας μην ξεχνάμε ότι η υδάτινη πόρη... η ίδια μας η τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουμε επηρεάζονται και αυτά από το ζήτημα της μικροβιακής αντοχής. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα αυτή νομοθεσία, κάθε γεωργική εκμετάλλευση θα πρέπει να ακολουθεί τις βασικές αρχές της υγείας των ζώων και θα πρέπει να χρησιμοποιεί πολύ συντηρητικά, πολύ προσεκτικά τα λεγόμενα EVMP τα κτηνιατρικά φάρμακα. Η νομοθεσία αυτή θα είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό το ότι καταφέραμε αυτή τη στιγμή να καταλήξουμε σε ένα πολύ σαφή κανονισμό, έτσι ώστε ακόμα και όταν μιλάμε για μια γελάδα, για ένα χείρο ή για ένα δέσποτο σκύλο, οι συστάσει είναι παντού οι ίδιε. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε ταλαιπωρία του ζώου, οποιαδήποτε καταπώνηση του ζώου, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται. Ένα κεντρικό επίση σημείο τη νέα νομοθεσία είναι ότι θα πρέπει να εκπονηθεί ένα κατάλογο μεταδοτικών ζωικών νόσων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Όπω για παράδειγμα οι ασθένειε που επηρεάζουν μια γεωργική εκμετάλλευση και το καθεξής. Και αυτό συνάδει και με τα πρώτα τμήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Το γεγονός ότι θα καταρτιστεί ένας τέτοιος κατάλογος είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και θα γίνει μέσω πράξεων κατεξοδότηση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα από αυτού. Πραγματικά θεωρώ ότι τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά. Είχαμε στο παρελθόν για 50 χρόνια 39 διαφορετικές οδηγίες και κανονισμούς και επιτέλους, επιτέλους όλα αυτά θα αντικατασταθούν από έναν και μοναδικό ξεκάθαρο νόμο, από έναν κρυστάλλινο κανονισμό, ο οποίος θα είναι εύληπτος, τουλάχιστον για τα 25 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σε καθημερινή βάση θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτόν τον κανονισμό. Συνεπώς, νομίζω ότι μέσω του κανονισμού αυτού δίνουμε ένα πάρα πολύ θετικό παράδειγμα ότι μπορούμε να πετύχουμε δηλαδή τους στόχους της Επιτροπής Juncker, να έχουμε δηλαδή μία αποσαφήνιση των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρους κανονισμούς, ξεκάθαρες οδηγίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 10 Ιουνίου η Κορεπέρα επιβεβαίωσε την υποστήριξη για την συμφωνία αυτή στην οποία έχουμε καταλήξει με το Συμβούλιο και ελπίζω τώρα πραγματικά ότι όλοι οι συνάδελφοι θα υπερψηφίσουν την πρόταση αυτή όπως ακριβώς έκανε και το Συμβούλιο στις 10 Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε να σας ε, συγχαρούμε για πρώτη φορά ο κύριο Ντάφμαν ε, θα έχει το λόγο. Παρακαλώ μην μιλήσετε περισσότερο από 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, κατ' ουσίαν θέλω να φέρσω μόνο την κυρία Πάουλσεν η οποία έβαλε σε αυτό τον τριμερή ε, διάλογο την ψυχή της, έβαλε τα πάντα, τα έδωσε όλα. Ε, θέλω λοιπόν να πω ότι ε, εντάξει πραγματικά την ευχαριστώ πάρα πολύ και σε τελική ανάλυση, μην ξεχνάτε, βρήκαμε μια λύση. Δεν χρειάζεται βέβαια να μπω σε λεπτομέρειε γιατί συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η κυρία Πάουλσεν. Καταλήξαμε σε μια λύση που είναι πολύ κοντά στην διαπραγματευτική εντολή που είχε δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός ο τριμερής διάλογος πράγματι οδήγησε ε, στο να έχουμε τελικά ένα πολύ λογικό ε, κανονισμό σχετικά με την ε, υγεία των ζώων και σχετικά με τις ε, μεταδοτικές νόσους. Τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μου την πολιτική ομάδα, με άνεση θα ψηφίσουμε αύριο, κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σμιτ έχει το λόγο. Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομο. Θα συγχαρώ την κυρία Πάρσεν Πάντοτε συγχαίρουμε τους εισηγητές μας, αλλά το εννοούμε αυτή τη φορά. Η κυρία Πόλσον πραγματικά έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για ένα πολύπλοκο ζήτημα. Και νομίζω ότι χάρη στην κυρία Πόλσον, στην ομάδα της και τη γραμματεία, είχαμε αυτή την τόση, το τόσο καλό αποτέλεσμα. 50 είναι τα εφτάμενα κείμενα που προσπαθούν ε, να επηρεάσουν τις ζωές των 20 εκατομμύρων ανθρώπων που εργάζονται ε, στον τομέα της ακτινοτροφίας. Ενώνονται λοιπόν αυτοί 50 σε έναν κανονισμό συνεκτικό. Σίγουρα θέλουμε την υγεία των ζώων να την ε, συνδυάσουμε και με την ε, καλή μεταχείρισή τους. Θέλουμε διευκρινήσεις από την Κομισιόν για το πώς θα προχωρήσει σε κάποια ζητήματα. Συγχαρητήρια όμως από την ομάδα μας, την κυρία Πάρσο και θα στηρίξουμε το πακέτο. Ευχαριστώ πολύ. Το ζήτημα της υγείας των ζώων είναι πολύ σημαντικό από ό,τι μπορεί να φαντάζονται ορισμένοι, γιατί έχει άμεση σχέση με την ανθρώπινη υγεία, την οτροφία, ο τρόπος με τον οποίο εκτρέφονται ή αντιμετωπίζονται θεραπευτικά τα ζώα είναι σημαντικός. Ε, δεν πρέπει να κάνουμε ε, τυχαία πράγματα, ιδίω ε, με τη βιομηχανική κτηνοτροφία. Ξέρετε ότι φανέρωσε ο τύπος ε, εξ ε, πολύ κακές πρακτικέ στον τομέα της κτηνοτροφίας. Λόγω του φιλελεύθερου συστήματος υπάρχουν κάποιες αποκλήσεις. Δεν θα πρέπει όμως ούτε την υπερβολική χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων να τη συνδέσουμε με την ανάγκη για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην κτηνοτροφία. Jutro odbędzie się głosowanie. Po tych wypowiedziach będzie głosowanie. Τελείωσε τώρα ο κατάλογος των αγοριτών. Ε, μία ψηφοφορία θα λάβει η χώρα και μετά ε, το θέμα θα το παραπέμψουμε στην Προεδρία. Κύριε Σανιό, είχα ζητήσει και εγώ να μιλήσω κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, Όσον αφορά την ε, διανομή των ε, φαρμάκων, αυτό είναι πιο εύκολο από αυτά που συζητάγαμε πριν. Ε, στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αλλά ξέρετε κάτι, θέλω η Επιτροπή να με ενημερώσει. Γιατί έχω γράψει εδώ σημειώσει μου ότι η Κομισιόν θα ήθελε τα κράτη-μέλη να οργανώσουν δυνατότητες διανομής φαρμάκων. Σας είπα, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν αυτοί οι ειδικοί για θέματα κτηνιατρικά, γίνεται λόγο στην έκθεση της κ. Πάουλσεν για την διανομή των φαρμάκων. Συγγνώμη, συγγνώμη, τα, έκανα, τα μπέρδεψα. Ε, κοιτάξτε πράγματι, τα μπερδέψατε, μιλήσατε για το επόμενο θέμα. Λοιπόν, εσείς θέλετε να μιλήσετε για τα κτηνέτρικα φάρμακα, αυτό είναι το έξι. Τώρα, εγώ πάω πίσω. Ε, πάμε ε, να πούμε ότι το θέμα θα παραπεμφθεί στην Ολομέλεια, στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Πάουλσεν. Πάμε στο επόμενο θέμα και θέλω να σας ότι καταρχήν σε ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Θέλω να σας πω το εξής, ότι στην έκθεση της κυρία Αγγιλέδα η καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση τροπολογιών είναι 26 Ιουνίου, 12 η ώρα το μεσημέρι. Και τώρα πάμε στο σημείο υπαρθμών 6, κτηνιατρικά φάρμακα. Υπάρχει, αυτή είναι μια έκθεση της ε, Καθήλυνα Αρμόδιας Επιτροπής. Αρμόδια είναι Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και τώρα θα συζητήσουμε για τις τροπολογίες ε, στην, στο σχέδιο της ε, γνωμοδότησης θα μας παρουσιάσει το θέμα η κυρία Μαρίτ Πάουλσεν. Το θέμα αφορά τα κτηνιατρικά φάρμακα αρμόδια. Όπως σας είπα είναι Επιτροπή Ένδια. Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα με πάρα πολλές τροπολογίες που σημαίνει ότι είναι απαραίτητο στον τομέα αυτό ε, να απλουστευτεί η διαδικασία.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 σε σχέση με αυτό το πολύ σημαντικό κείμενο νομοθετικού περιεχομένου. Ίσως να είναι μια λεπτομέρεια, παρόλα αυτά έχει τη σημασία της στο πλαίσιο αυτού του τεράστιου πακέτου που εξετάζουμε. Συνολικά έχουν κατατεθεί 460 τροπολογίες. Αρχικά θεώρησα ότι είναι καλό αυτό. Δεν βλέπω να υπάρχουν ε, άλλα τα προβλήματα μίζωνας αντιπαραθέσεις. Σίγουρα υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες που εκφέρουν απόψεις και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί γιατί δεν μπορούμε να περιλαμβάνουμε απόψεις και γνώμες αν να πρόκειται για νομοθεσία. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε λοιπόν. και να παραμείνουμε στα γεγονότα σε στοιχεία. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το ίδιο θέλουμε, δηλαδή τη βελτίωση της πρόσβασης στα κτηνιατρικά φάρμακα. Θέλουμε να αναπτυχθεί ο τομέας, να είναι αποτελεσματικός και να αναλάβουμε επίσης αποτελεσματικά και με αποφασιστικότητα δράση κατά της μικροβιακής αντοχής. Ιδίω δε όταν μιλάμε για τη διαρροή των προϊόντων αυτών είτε στο έδαφο είτε στον υδροφόρο ορίζοντα. Πρέπει να συμφωνήσουμε πάνω σε μια σειρά από σημεία και να καταθέσουμε και συμβαστικές τροπολογίες. Για παράδειγμα, πρέπει να βρούμε μια λύση σε ένα ζήτημα το οποίο επανέρχεται, δηλαδή ποιος μπορεί ή έχει το δικαίωμα να συνταγογραφήσει ένα φάρμακο. Η άποψή μου είναι εξής. θα πρέπει να έχουμε έναν ειδικό που μπορεί να μην είναι κτηνίατρος, ο οποίος θα μπορεί να συνταγογραφεί φάρμακα μεν, τα οποία όμως όταν δεν συνταγογραφούνται από κτηνίατρο, να μην πολλούνται παρά μόνο στη χώρα όπου το λόγο άτομο θα έχει καταρτήσει τη συνταγή, δε αν υπάρχει διασυνοριακή πόλη στο φαρμάκου, η συνταγή θα πρέπει να γίνεται από κτηνίατρο, διαπιστευμένο. Όταν έχουμε συνταγή από έναν ειδικό, από έναν επαγγελματία του κλάδου της όμως δεν είναι κτηνίατρος, αυτή η συνταγή θα ισχύει μόνο στη χώρα η οποία αναγνωρίζει την ύπαρξη των λόγων επαγγελματία. Ε, κυρίως για το Ηνωμένο Βασίλειο ε, πρόκειται Εκεί υπάρχουν ε, επαγγελματίε στο τομέα τη που μπορούν να συνταγογραφούν παρότι όχι κτηνιατρικά φάρμακα. Το 2006 εγκρίθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νομοθέτημα για τα αντιβιωτικά. Δυνάμει του κειμένου αυτού τα αντιβιωτικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για το σκοπό της εκτροφής, της πενοτροφίας. Ήταν πολύ σημαντικό και είχαμε πει ότι η χρήση αντιβιωτικών θα μειωθεί με τον τρόπο αυτό. Δεν συνέβη αυτό. Η χρήση αντιβιωτικών συνέχισε να αυξάνεται, γιατί μιλούσαμε για προφύλαξη, προληπτική δηλαδή χρήση του φαρμάκου. Όμως είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιούνται τα κτηνιατρικά φάρμακα για την προληπτική αγωγή. Και τώρα περνάμε στην μεταπροφύλαξη. Δεν θα πρέπει και πρέπει να προσέξουμε για μια ακόμη φορά να έχουμε κάποιες υφαίες ζώνες σε ένα νομοθέτημα που θα επιτρέπει τελικά την παράκαμψη της νομοθεσίας και τη μη τήρηση των στόχων που έχουμε θέσει. Πρέπει να συμφωνήσουμε λοιπόν ως προς τους ορισμούς, ώστε να είναι η σαφέστερη δυνατή για την μεταφυλακτική χρήση κυρίως αντιβιωτικών. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πλέον λεπτό ζήτημα της νομοθεσίας για την χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων. Μεταφύλαξη λοιπόν η αγωγή ελέγχου. Έχουμε συμφωνήσει επί της αρχής ε, με τους Σκιώδης και θα δώσουμε στους εργάτες μας την δυνατότητα να εργαστούν και θα τα ξαναπούμε στο Στρασβούργο. Θα ήθελα να ακούσω τώρα τις δικές σας απόψεις, επαναλαμβάνοντας ότι αυτό που είναι σημαντικό κατά την άποψή μου, είναι να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μια νομοθεσία που δεν θα έχει υφαίες ζώνες. Για να μην συνεχίσουμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτη κυρία Σουσκάτ. Κύρια Πόλσεν, πράγματι ήταν χαρά για μένα να συνεργαστώ μαζί σας ε, και θέλω να πω ότι κατά την άποψή μου εμείς ως πράσινοι πιστεύουμε ότι το θέμα σχετίζεται άμεσα και με την φύση της ε, γεωργίας μας. Δεν πιστεύουμε ότι η βιομηχανική γεωργία εξυπηρετεί ε, τα ζώα μας και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα, τις φαρμακούχες ζωοτροφές ε, και να τις χορηγούμε στα ζώα μας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα καλυφθούν τα κενά σε όλα τα δεδομένα, κυρίως όσον αφορά την ε, αξιολόγηση περιβαλλοντικών ε, κινδύνων, να μην ζητάμε εγκρίσεις χωρίς περιορισμούς. Χρειαζόμαστε αυστηρότερους κανονισμούς για να περιορίσουμε την ε, κανονική χρήση των φαρμάκων, την καθημερινή, κυρίως ε, για ζώα ε, που δεν είναι άρρωστα. Αυτά τα προφύλαξη και μεταφύλαξη, αυτά είναι λιγάκι ύποπτα και εμείς αυτούς τους νέους ορισμούς τους βρίσκουμε πολύ περίεργους. Θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητο να κυκλοφορούν γιατί είναι απειλή για την δημόσια υγεία. Επίσης έχουμε καταθέσει τροπολογίες ε, για τις κατευθυντήρες γραμμέ σχετικά με την αντοχή στα αντιβιωτικά. Ε, κατά την άποψή μας ε, κάποια αντιβιωτικά θα πρέπει να προβλέπονται αποκλειστικά και μόνο για την υγεία των ανθρώπων. Προτείνουμε και ένα σύστημα μονογράφησης για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις από τη χρήση αντιβιωτικών όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα ζυζανιοκτώνα. Αυτό να γίνεται σε καθημερινή βάση έτσι ώστε να μπορούμε να αποκτήσουμε πληροφορίες για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία. Και όχι μόνο για τα ζώα τα οποία υποτίθεται ότι ε, τους επιβάλλεται μια θεραπεία με αντιβιωτικά. Να υπάρχουν καλύτερα στοιχεία όσον αφορά τα αντιβιωτικά, ε, την καλύτερη επαγρύπνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι και προσβλέπω στη συνέχιση των συζητήσεων. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλοι ομιλητέ παρακαλώ. Ο κύριος Αγνού, αλλά σας παρακαλώ πολύ να είστε σύντομος. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξαναπαίρνω τώρα το λόγο λίγο απότομα, αλλά βλέπουμε αυτή τη στιγμή... Θα ήθελα να ρωτήσω, αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή είτε στην έκθεση που έχουμε στο σημείο 4, στο σημείο 6. Σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μας πει αν τα SQPs αυτοί οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να συνεχίσουν να χορηγούν κτηνιατρικά φάρμακα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καταλαβαίνω ότι εσείς μας λέτε ότι μπορούμε να έχουμε αυτούς τους ε, ανθρώπους, αλλά θα ήθελα μια ξεκάθαρη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τους ανέχεστε απλώς ή μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται στο, στο Βασίλειο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιούσο. Θέλω να συγχαρώ καταρχάς την κυρία Πάλσεν για την εξαιρετική της δουλειά όπως βέβαια κάνει όποτε λαμβάνει ένα ζήτημα, ιδίω αν σχετίζεται με την υγεία των ζώων. Έχω καταθέσει αρκετέ τροπολογίε για την έκθεση, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ γενικά στα σημαντικότερα ζητήματα στι σημαντικότερε τροπολογίε, από τι οποίε κάποιε αναφέρονται στη διαθεσιμότητα των κτηνιατρικών φαρμάκων, γιατί πραγματικά χρειάζονται φάρμακα για ίσονε χρήσει ή για είδη ίσονο σημασία και έχω καταθέσει σχετική τροπολογία για να υπάρχει διαθεσιμότητα των εν λόγω φαρμάκων. Επίση, είναι σημαντικό, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, στον κανονισμό αυτό να μιλάμε για τις λεγόμενες διαδοχικές συνταχογραφήσεις ε, που περιλαμβάνεται στην οδηγία του 2001 ώστε σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κτηνιατρικά φάρμακα για ένα συγκεκριμένο είδος ή για μια συγκεκριμένη νόσο, ο κτηνίατρος, ο αρμόδιος κτηνίατρος, πάντων ο αρμόδιος για την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, στη χώρα μου πρόκειται πάντα για κτηνίατρο, να μπορεί να συνταγογραφήσει φάρμακα που προέρχονται για ανθρώπινη χρήση. Και στι τροπολογίε μου έχω συμπεριλάβει κατά λέξη αυτό που λέει η οδηγία ε, του 2001 Επίσης, ό,τι αφορά ε, τη χρήση κοινωτικών φαρμάκων που είχαν πρώτερη έγκριση και δεν ε, ήταν στην αγορά ενός κράτους μέλους για τρία χρόνια, ε, έπαβε να ισχύει αυτή η έγκριση αυτή τη κυκλοφορία. Αυτό ήταν ίσχυε για χρόνια στην νομοθεσία και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να ισχύει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση, τα συστήματα ε, δεν θα πρέπει να είναι ισοδύναμα με τις περιοδικές εκθέσεις ασφάλειας. Αυτές οι ασθενείς λέει ομιλήτρια πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν και τα στοιχεία προφανώς εννοεί για να μπορούμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τη συντάκτρια της έκθεσης εγώ νομίζω ότι όλα αυτά αποτελούν μια πολύ καλή βάση, πολύ καλή έκθεση. Θα βασιστούμε σε αυτή. Εγώ έχω, ή έχω ήδη καταθέσει κάποιες ε, τροπολογίες και πολλά από αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως ε, για τις ε, φαρμακούχες ζωοτροφές ή αυτά που είπαμε για τους ορισμούς, πώς θα ορίσουμε τα αντιβιωτικά, ορισμός της προφύλαξης, της μεταφύλαξης, της θεραπείας. Για όλα αυτά θα υπάρξει μια ικανοποιητική λύση. Υπάρχει ένα θέμα που εγώ θέλω να θίξω, δηλαδή ε, έχω κυρία Πόλσεν λιγάκι την εντύπωση ότι αμφισβητείται λιγάκι το, την, την ιατρική διανομή και αυτό το κάνετε με τις ε, τροπολογίες Εγώ δεν θα προχωρούσα τόσο πολύ Νομίζω ότι αυτό αποδείχθηκε αρκετά αποτελεσματικό για να περιοριστεί η χρήση των αντιβιωτικών. Πολτσακ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί συμφωνώ με πολλούς συναδέλφους. Νομίζω ένα βασικό ερώτημα αφορά στην ε, ε, διάρκεια, στη χρονική διάρκεια της προστασίας δεδομένων. Αυτή είναι μια πολιτική συζήτηση και είναι σαφές ότι ισχύοντες κανονισμοί για την ε, κτηνιατρική αγωγή είναι μικρής διάρκειας. Αν επεκταθεί η διάρκεια αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα περιοριστούν τα γενώσιμα που έχουν τη μισή τιμή των ε, πρωτότυπων φαρμάκων. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω τους κινδύνους ε, που μπορούν να προκύψουν αν δεν υπάρχουν πρωτότυπα φάρμακα δεν μπορούν να υπάρχουν και γενώσιμα. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε λιγάκι για ποιο χρονικό διάστημα ισχύει η προστασία ε, και από αυτού συμφωνούν και ορισμένοι παραγωγή γενοσύμων. Και όλα αυτά πρέπει να είναι και υπό τον έλεγχο του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Και όσον αφορά την διανομή από το διαδίκτυο, υπάρχει απαγόρευση διακίνησης συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Σωστό αυτό. Όμως τα μη συνταγογραφούμενα θα πρέπει να είναι δυνατόν να πολλούνται μέσω διαδικτύου. Εγώ θα ήθελα να φερθώ και στο θέμα ε, του κτηνιάτρου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριο Σφεγό. Βλέπουμε σήμερα ότι έχουμε τη σύσταση μιας νέας πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως, μπορείτε πλέον να αποφεληθείτε από τους νέους αυτούς ευρωβουλευτές με τις νέες πιο ενισχυμένες αρμοδιότητες. Όσον αφορά τώρα τα κτηνιατρικά φάρμακα. Νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να έχουμε απελευθέρωση τη διακίνηση των ε, φαρμάκων αυτών, ιδίω των στεγογραφούμενων. Και ιδίω δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την πώληση μέσω διαδικτύου. Είναι πολύ σημαντικό κάθε κράτος μέλος να μπορεί να έχει την απόλυτη διαχείριση του ποιο θα μπορεί να συνταγογραφεί τα φάρμακα αυτά και αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο τότε νομίζω ότι το κείμενο αυτό θα οδηγήσει τελικά στην ε, παραποίηση και την παράνομη διακίνηση των φαρμάκων αυτών. Στην αντίθεση με τόσα λέει η συγγήτρια στο κείμενό της, οι κτηνίατροι δεν κάνουν την ίδια δουλειά με τους ιατρούς. Δεν υπάρχει, όπως γνωρίζετε για τα ζώα, ούτε κάλυψη από κάποιο ταμείο, ούτε η ιατροφαρμακευτική ασφάλιση. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο οι κτηνοτρόφους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν θα πρέπει σε κανένα περίπτωση να αυξήσουμε όλο και περισσότερο τις τιμέ τέτοιων υπηρεσιών που είναι ήδη πολύ ψηλές και πλήττουν πάρα πολύ τον κτηνοτροφικό κλάδο. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί για τα σημεία αυτά, στα σημεία αυτά το προτινόμενο κείμενο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο σκιώδης ηγητής τώρα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, όσον αφορά αυτήν την έκθεση, νομίζω πρέπει να θεωρούμε ότι η έκθεση αυτή πρέπει να είναι ρεαλιστική. Ρεαλιστική όσον αφορά τις δραστηριότητές μας. Δεν μπορεί κανείς την έκθεση να την περιορίσει μόνο στα αντιβιωτικά. Εδώ μιλάμε για τη γεωργία, για την αλία και υπάρχουν κάποιοι κανόνες ε, που ισχύουν και για την υγεία των ζώων. Έχουμε εντατική γεωργία, μαζική κτηνοτροφία, όπου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κάποιες ουσίες που αναφέρθηκαν σήμερα εδώ. Εξάλλου, την έκθεση για την χορήγηση φαρμακούχων ζωοτροφών, ε, θα πρέπει να έχουμε κατά νου την πραγματικότητα και να μην θεωρήσουμε ότι αυτό είναι εργαλείο για να χορηγούνται απλά αντιβιωτικά. Η έκθεση είναι πολύ πιο ευρεία και περίπλοκη. Κατ' ουσίαν πρόκειται για την πρόσβαση στα φάρμακα που κατά την άποψή μου είναι ε, πολύ σημαντική και αυτό πρέπει να γίνεται μέσα από ένα κεντρικό μητρό έτσι ώστε να μην βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου οι πολυεθνικές απλά θα επιβάλλουν τη γνώμη τους και εμείς απλά δεν θα έχουμε πρόσβαση σε κάποια φάρμακα. Τώρα, όσον αφορά την φαρμακοεπαγρύπνηση, ε, θα πρέπει να εισαχθεί η, εφα... φαρμακοεπαγρύπνηση με ελέγχους βέβαια και περιοδικούς ελέγχους. Νομίζω ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός είναι πολύ σημαντικός, όπως είναι εξίσου σημαντικό να ελέγχουμε και την χρήση των αντιβιωτικών και των φαρμάκων φάρμακα χορηγούνται πολύ περισσότερο από αντιβιωτικά. Μπορούμε να περιορίσουμε τα αντιβιωτικά ε, για πρόληψη, για προληπτικούς λόγους και λόγους ε, προφύλαξης. Και με τον τρόπο αυτό ε, μπορούμε να περιορίσουμε και το κόστος. Βεβαίω όλα αυτά πρέπει κανένα τα ελέγχει, να ελέγχεται και η πώληση από το διαδίκτυο και κάτι τελευταίο που έχει σχέση με την καινοτομία. Έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες ε, προσπαθούν να επεκτείνουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες και πρέπει να μεριμνήσουμε να υπάρχει σωστή ενημέρωση και τα φάρμακα να ε, είναι ανταγωνιστικά, να παραμένουν ανταγωνιστικά για τους ε, κατασκευαστές. Και κάτι άλλο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε η δική μας Επιτροπή να μην κατακυδεμονευτεί από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. μισή λεπτά μιλήσατε εσείς. Η κυρία Μούλερ έχει το λόγο. Ähm, ich habe Müller verstanden. Müller Εγώ δεν λέγομαι Müller. Μίλλερ κατάλαβα. Μίλιο λέγομαι παρακαλώ. Λοιπόν, έχω να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Ε, καταρχήν θέλουμε στην κυρία Πάουλσε. Νομίζω όμως ότι όσον αφορά την χρήση των αντιβιωτικών, κυρίως όσον αφορά τα ε, αντιβιωτικά ρεζέρβα, ε, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε να βρούμε κάποιες λύσεις. Όσον αφορά λοιπόν τα εφεντρικά αντιβιωτικά, νομίζω ότι ε, θα πρέπει λιγάκι να το εξετάσουμε αυτό και μάλιστα ε, να πούμε ότι αν υπάρξουν ε, ε, κάποια ευρήματα θα πρέπει να αντιδράσουμε. Όσον αφορά την χρήση γενικότερα των κτηνιάτρων και την ε, ε, γενικότερη δραστηριοποίησή τους. Θα πρέπει να το διατηρήσουμε αυτό για να μην συμβαίνει αυτό που ήδη συμβαίνει. Δηλαδή να χρησιμοποιούνται τα αντιβιωτικά όχι ως ε, μέσα αγωγής και θεραπείας αλλά ως προφυλακτικά μέτρα. Η κυρία Αγγιλέρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Συμφωνώ με ορισμένα από όσα επισήμανε η κυρία Γιούσο. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να λησμονούμε τις δυσκολίες που συνεπάγεται η πρόσβαση ε, σε φάρμακα για τα είδη ίσονος σημασίας. Όταν ολοκλήρωσε η σα είπε ότι πρέπει να περιορίσουμε να έχουμε μια περιορισμένη χρήση, είπε, των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην προληπτική αγωγή. Συμφωνώ. Όμως το πρόβλημα είναι η διαθεσιμότητα φαρμάκων για τα είδη ίσονα σημασία. Πώ θα λύσουμε το πρόβλημα αυτό, Εγώ δεν έχω τη λύση βέβαια, αλλά θέτω το ζήτημα. η εκτίμηση που κάνατε και το ότι επιμένετε στο να ακολουθήσουμε τις βέλτιστες κτηνιατρικές και νοτροφικές πρακτικές είναι σημαντικό. Γίνονται πολλά. Ο κ. Φέντριλε πριν επέμεινε ότι σε ορισμένες χώρες ήδη γίνονται νέα πράγματα, ενδιαφέροντα, αλλά θα πρέπει να διατηρήσουμε την διαφορετικότητα, την πυκλομορφία της Ευρώπης. Πολλά μπορούμε να το μηγενοποιήσουμε, αλλά το κλίμα, και κάποιες άλλες συνδίκες και προϋποθέσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αν και συμφωνώ με αυτό το στόχο που θέσατε. Και κάτι τελευταίο κύριε Πρόεδρε, ξέρω ότι τελειώνει ο χρόνος μου, κατάργηση των διαδοχικών συνταγογραφήσεων. Και αυτό με, με ανησυχεί και εμένα, όπως το είπε και η κυρία Αγιούσο. Grazie, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να συγχαρώ την συνάδελφο Πάουελσεν και κατάφερα και εγώ να συμβάλλω μέσω παρατηρήσεων ως σκιώδης εισηγητής. Ξέρετε ότι έχουμε 460 τροπολογίες, ε, έπρεπε να βρούμε ένα κάποιο συμβιβασμό, έτσι δεν είναι, για να καταλήξουμε σε ένα εύληπτο καλό κείμενο. Θα ήθελα τώρα να επικεντρωθώ σε κάποια σημεία τα οποία έχουν ήδη θίξει ορισμένοι συνάδελφοι. Πρώτον, η χρήση των αντιβιωτικών. Σε κοινοτικό επίπεδο, όπως υπόθηκε, δεν έχουμε συγκεκριμένα επιστημονικά δεδομένα προκειμένου να γνωρίζουμε αν τελικά έχουμε σωστά μέτρα και αν τελικά έχουμε οδηγηθεί στο φαινόμενο αυτό της μικροβιακής αντοχής. Χρειαζόμαστε λοιπόν συγκεκριμένα δεδομένα και καλύτερη συλλογή των δεδομένων όσον αφορά τη χρήση των ίδιων των αντιβιωτικών για να έχουμε μια καλύτερη παρακολούθηση της χρήσης τους. Ένα άλλο σημαντικό σημείο στην έκθεση αυτή είναι το να καταφέρουμε να διευκρινίσουμε ακριβώς, υπόθηκε άλλωστε και αυτό, ποιος ήταν ο, ο ρόλος των ίδιων των κτηνιάτρων. Ξέρετε ότι δίστανται οι απόψεις, εγώ από προσωπικής πλευράς έχω κάποιες αμφιβολίες, είμαι λίγο επιφυλακτικός για το αν θα μπορούσαν τελικά οι κτηνίατροι να χορηγούν και μάλιστα να πουλούν και αντιβιωτικά φάρμακα. Νομίζω ότι πρέπει και αυτό κάπως να το τονίσουμε στην έκθεση και να ρυθμίσουμε καλύτερα το ρόλο τους. Τα υπόλοιπα σημεία που θέλω να θίξω είναι πρώτον να καταφέρουμε να αναφέρουμε το ζήτημα της φάρμακοεπαγρύπνησης. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να παρακολουθούμε και την παρουσία κάποιων καταλήπων από αντιβιωτικά στους υδροφόρους ορίζοντες ή στο ίδιο το έδαφος. Έπειτα έχουμε και το ζήτημα της online πώληση, της πώληση στο διαδίκτυο και αυτό πρέπει να το ρυθμίσουμε, διότι όπως υπόθηκε και από τον προλαλήσαντα, έχουμε σαφώς όσους λένε ότι θα πρέπει να απαγορέψουμε τέτοια πώληση, ενδεχομένως ναι, αλλά από την άλλη ακόμα και αν δεν απαγορέψουμε την πώληση αυτή, θα πρέπει να έχουμε ένα πάρα πολύ αυστηρό έλεγχο για την πώληση και τη διακίνησή τους. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να καταφέρουμε μέσα στο κείμενο αυτό να συμπεριλάβουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την κυρία Πάουλσεν για την πολύ καλή της γνωμοδότηση. Είχαμε όντως μια πολύ καλή συνεργασία. Να επανέλθω στο ζήτημα της αδειοδότησης και μάλιστα υπέβαλα και σχετική τροπολογία. Υπέβαλα λοιπόν μια τροπολογία προκειμένου να είναι δυνατό να δίδεται μια αποκεντρωμένη αδειοδότηση. Δηλαδή δεν ζητώ εδώ πέρα μια νέα διαδικασία, αλλά την δυνατότητα να τροποποιηθεί η φυστάμενη διαδικασία και να έχουμε μια αποκεντρωμένη αδειοδότηση για τα φάρμακα αυτά. Νομίζω ότι αυτό θα διευκολύνει κάπως τα πράγματα. Σας ζητώ να υποστηρίξετε λοιπόν αυτή την τροπολογία και περιμένω να δω πώς θα εξελιχθούν οι συζητήσεις την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φέντερλε έχει το λόγο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή έκθεση ε, και είναι ε, σαφές ότι εδώ αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στα αντιβιωτικά. Αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε σοβαρά όλα τα φάρμακα, γιατί όπως ελέγχθηκε προηγουμένως, ε, δεν είναι ότι όταν χρησιμοποιούνται αντιβιωτικά για ασθένειες προκαλείται αντοχή. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που οι γιατροί καλούνται να δείξουν κάποια υπευθυνότητα. Ε, να ελέγχουμε τη χρήση των αντιβιωτικών γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό ε, θα φτάσουμε στην ε, θεραπεία που υπήρχε πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό λοιπόν θα σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα για την υγεία. Η κυρία Πόλσεν είχε μια πολύ σημαντική συνεισφορά ε, στην Σουηδία ξεκινήσαμε πολύ πιο παλιά. Ε, τα αποτελέσματα είναι τα ίδια, έστω και εδώ ήταν αρκετά ε, πρόσφατη η κίνηση. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει η ίδια πούληση στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπάρχουν τρία θέματα που θέλω να δείξω. Το ένα θέμα είναι αυτό το ε, δικαίωμα άσκηση επαγγέλματος ε, για τους εκτινέατους. Είναι σημαντικό αυτοί να μπορούν να συνταγογραφούν φάρμακα. Αυτό συνηθίζεται στη Γερμανία. Και πρέπει να δει κανεί και το δεύτερο θέμα τη όλη υπόθεση, ότι δηλαδή στην περίπτωση που χορηγεί φάρμακο ιατρό, αναλαμβάνει και την ευθύνη. Αυτά πάνε από μαζί, από κοινού. Γιατί αλλιώ τι γίνεται, μοιράζουμε τις ε, ευθύνε, αρμοδιότητες, ο ένας γράφει, ο πουλάει, ο αγοράζει και όταν συμβεί κάτι πολύ, κανείς δεν είναι, όταν συμβεί κάτι, κανείς δεν είναι υπεύθυνο. Κατά τα άλλα, ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί το ποιο θα συνταγογραφεί, γιατί πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Και όσον αφορά τα εφεδρικά αντιβιωτικά, θα πρέπει να βρούμε μια πολύ αξιόπιστη ε, περιοριστική λύση η οποία θα μπορεί και να αντέξει στη δημόσια συζήτηση. Κύριε Ντές, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να πω μερικά πράγματα ε, σχετικά με αυτά που ελέγξαν για τα αντιβιωτικά. Στη Γερμανία Υπάρχει Ινστιτούτο Προστασίας ε, Καταναλωτή και Ψηφιστικής Βοήθειας και εκεί αναφέρεται το 2013 μόνο το 1% ε, του συνόλου ε, των αντιβιωτικών που πουλήθηκαν ήταν κτηνιατρικά ενώ το ποσοστό στην ανθρώπινη χορήγηση το αντίστοιχο ποσό ανέκτησε στο περίπου 17%. Άρα δηλαδή όταν πρόκειται για αντοχή στα αντιβιωτικά εδώ δεν φταίει η κτηνιατρική και τα κτηνιατρικά φάρμακα αλλά όπως σας είπα αυτό το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο καταλήγει στο ότι και στα νοσοκομεία ε, υπάρχουν καταστάσεις που πρέπει να αλλάξουν. Δεν μπορεί κανείς ο καθένας να μπαίνει έτσι χωρίς λόγο ε, στο νοσοκομείο. Έτσι από τον δρόμο ανοίγει την πόρτα και μπαίνει. Μπορεί να μεταφέρει αντιβιωτικά, συγγνώμη, συγχωρείτε, ε, μικρόβια τα οποία κατόπιν διαδίδονται μέσα στο νοσοκομείο και προκαλούν πρόβλημα. Πολύ ωραία λοιπόν, λέει ο πρόεδρος, έκλεισε η συζήτηση. Ε, και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ζαρό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν να ε, περάσω στην ουσία, θα ήθελα όπως και όλοι όσοι έλαβαν το λόγο να συγχαρώ και εγώ την κυρία Πόλσεν για το εξαιρετικό της έργο. Η συνεργασία μαζί ήταν πραγματικά χαρά μας και προσωπική χαρά για εμένα, αν μου επιτρέπετε. Υπάρχουν κάποια σημεία από των οποίων θα ήθελα να πω δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα, ορισμός προφύλαξης, δηλαδή προληπτικής αγωγής, μεταφύλαξης, δηλαδή αγωγής ελέγχου κτλ. Ήρθαμε σε επαφή με διάφορους φορείς, μιλήσαμε και με το Συμβούλιο και πρόσφατα μιλήσαμε και για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εκτινιάτρων που προέβαλε κάποια επιχειρήματα τα οποία νομίζω ότι αξίζουν την προσοχή μας ό,τι αφορά την εγκυρότητα των αδειών κυκλοφορίας πρόταση πεντέτους ανανέωσης θα το εξετάσουμε σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης, έγκρισης υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που δεν θα περάσει η έγκριση κάποιων φαρμάκων συγκεκριμένα από την κεντρική διαδικασία ιδίω για νέε δραστικέ ουσίε όπω συμβαίνει σήμερα, εμεί νομίζουμε ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να ακολουθείται η κεντρική διαδικασία. Πρώτον, για λόγους διαθεσιμότητας και δεύτερον, γιατί θα πρέπει να αξιολογηθεί το φάρμακο από τους ε, καλύτερους επιστήμονες και ειδικού από των κρατών μελών. Τώρα το όλο κεφάλαιο διαφοροποίησης προτείνεται να αντικατασταθεί από μια έκθεση αξιολόγησης της λειτουργίας ε, του κανονισμού του 2008. Ε, τα variations ε, κάνουμε συγκεκριμένα την ανάλυση, τη μελέτη αντικτύπους. Ό,τι αφορά την πρόταση τεχνικών εγγράφων, μια φορά και έναν καιρό το λέγαμε προστασία δεδομένων. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ισορροπία για να έχουμε από τη μία πρόθεση των επενδύσεων και προστασία του ανταγωνισμού αφετέρου. Έχουμε στοιχεία και το βλέπουν όλοι πιστεύω, δεν γυμνώ φθάλμου, ότι δεν έχουμε αρκετές δοκιμές για τα ζώα, ιδίως για είδη ισονοσημασίας και ιδίως για τα μικρά κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε, να πιέσουμε λίγο τον κλάδο με επενδύσει σε τομείς όπως για παράδειγμα είναι η μέληση μου έρχεται στο μυαλό. Ήταν αντιδυτικά για παράδειγμα αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διατηρήσουμε και τον ανταγωνισμό σε καλά επίπεδα. Να μην παράσχουμε μία ανεφόρο προστασία, ε, όπως ανέφερε κάποιος, ε, για τις αντιμικροβιακές ουσίες. Αυτό είναι βασική ανησυχία και όχι μόνη βέβαια, πολύ σωστά. Μεταξύ άλλων το είπε και ο κύριος Βιέγκας. Και μας οδήγησε να προτείνουμε την αναθεώρηση του, του ρυθμιστικού πλαισίου που σήμερα μπορεί και να με αναφέρει τίποτα για τις αντιμικροβιακές ουσίες και την αντιμικροβιακή αντοχή, η Κομισιόν προτείνει τουλάχιστον 15 νέες εντελώ ε, απαιτήσει από την υποχρεωτική στατιστική συλλογή δεδομένων για την ε, πώληση και χρήση αντιμικροβιακών ουσιών έως την δυνατότητα κάποια ε, σημαντικά αντιμικροβιακά ε, να χρησιμοποιούνται μόνο για τον άνθρωπο βάσει επιστημονικών ε, στοιχείων. Εμείς θα εξετάσουμε οποιαδήποτε υπόδειξη και σύσταση. Έχει ως στόχο την πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της ε, αντοχής στα αντιβιωτικά και αντιμικροβιακά, βέβαια με μέλημά μας πάντα την προστασία της υγείας ανθρώπου και, του, των ζώων. Φάρμακο, επαγρύπνηση. Δεν συμφωνούμε ότι έχουμε κάπως ε, μετριάσει τις διατάξεις. Βασιζόμαστε σε αιτήσιες εκθέσεις. Το 98% αφήνω τελώ. Το 98% αφήνουμε άθικτο, αλλά προτείνουμε να περάσουμε σε ένα σύστημα που θα παρακολουθεί συνεχώ όλες τι ανεκτήμητε ενέργειες όλων των κτηνιατρικών φαρμάκων. Μια προσέγγιση βασισμένη στους κινδύνους υιοθετούμε μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων που συμμετείχε ενεργά στη σύνταξη των διατάξεων αυτών. Πιστεύουμε λοιπόν και εμείς και ο ΕΟΦ ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την καλύτερη προστασία της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, για τις ε, online πωλήσει. Δύο-τρία δευτερόλεπτα για να σας εξηγήσω τι ακριβώς θέλουμε. Δεν πιστεύουμε ότι με τον κανονισμό, με τον ευρωπαϊκό κανονισμό μπορούμε να ξεφορτωθούμε με τη μία ε, την πώληση πλαστών ψευδοφαρμάκων από άλλες χώρες του κόσμου σε πελάτες που μπορεί να γνωρίζουν, μπορεί όμως και να μην γνωρίζουν τι αγοράζουν. Το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα, πριν από τέσσερα χρόνια. Στο πλαίσιο της οδηγίας ε, της έγκρισης παραπημένων ψευδών φαρμάκων, πλαστών φαρμάκων. Και ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό που θα επιτρέπει την αναγνώριση, την ταυτοποίηση αυτών των φορέων που είναι εγκεκριμένοι σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη-μέλη για να πωλούν online φάρμακα. Διότι αυτά τα φάρμακα σήμερα πολλούνται στην Ευρώπη. Εγώ δεν προτείνω να αλλάξει αυτό από εξουσιοδοτημένου πολιτέ. σε εθνικό επίπεδο. Μπορεί να είναι ε, φαρμακοποιοί, κτηνίατροι, σε ορισμένε περιπτώσεις. Ε, αν τα κράτη-μέλη, δεν θέλουν να αλλάξει αρχή. Θέλουν αυτό να περιλαμβάνει όλα τα μη συνταγογραφούμενα ή κάτι άλλο. Εμείς λέμε ότι τα κράτη-μέλη όταν εξουσιαστούν σε κάποιον να πουλήσει φάρμακα ε, online, λέει το άρθρο 107 συγκεκριμένα, μπορεί να το κάνει το κράτος μέλος, αφού βέβαια τηρούνται οι διατάξεις για την προστασία της δημόσιας υγείας. Άρα υπάρχει δυνατότητα επιβολής κάποιων περιορισμών από τα κράτη-μέλη. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να έχουμε μια σαφή διάταξη μια μάλλον σαφή δέσμη διατάξεων, ώστε οι εγκεκριμένοι ανοπολιτέ ε, να είναι νόμιμοι, να έχουν δηλαδή πραγματικά εξουσιοδότηση και έγκριση σε εθνικό επίπεδο για να πολλούν φάρμακα. Και έχουμε ένα template, το ίδιο ακριβώς ε, που είχαμε στην οδηγία για τα πλαστά ή παραπημένα φάρμακα για ανθρώπινη κατανάλωση, ανθρώπινη χρήση. Το τελευταίο είναι οι ερωτήσει των κυρίων Άγγιν και Φερό. Ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή τη αφήνει την κατάσταση ως έχει. Για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Νορβηγία υπάρχει μια ιδιαίτερη περίπτωση και εκεί λέμε τα άτομα που εξοδοτούνται να συνταγογραφούν εκτελετρικά φάρμακα σύμφωνα με τις ισχύωσε εθνικές διατάξεις. Τα επαγγέλματα, παραλαμβάνω, ε, ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο και τα προσόντα. Σε εθνικό επίπεδο δεν θέλουμε να παρέμβουμε και δεν έχουμε και κάποιο στοιχείο ότι υπάρχει πρόβλημα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στον τομέα των επαγγελματιών του κλάδου της υγείας των ζώων, κτηνιάτρους κτλ. Μιλάμε για τα φάρμακα την πληροφόρηση σήμερα. Δεν αλλάζει αυτή η αρχή. Νομίζω ήμουν σαφή, κύριε Άγγνιο, Ελπίζω τουλάχιστον. This is the commission proposal. Και βέβαια αυτή είναι η πρόταση τη Κομισιόν. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, εισηγείται, έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις παρατηρήσεις και για τις αντιδράσεις, αντιρρήσεις που είχατε. Προφανώς θα συνεχίσουμε τη συζήτηση που ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε και τις διαπραγματεύσει προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα σεβιβασμό. Είμαι πραγματικά πεπισμένη ότι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε επιτυχώς το έργο μας και θα είμαστε έστω κατά 90% όλοι ικανοποιημένοι. Είμαστε η Επιτροπή Γεωργίας, άρα η υποχρέωσή μας είναι να συνταχθούμε με τους αγρότες, με τους γεωργούς, με τους κτηνοτρόφους, να δούμε πώς έχει στην πράξη δραστηριότητά τους. Εγώ κοίταξα πάρα πολλές πρόσφατες έρευνες όσον αφορά την μικροβιακή αντοχή και ποιες είναι οι επιπτώσεις του φαινομένου αυτού στους υδάτινους πόρους, γιατί γενικότερα για τη ζωή στον πλανήτη μας. Και νομίζω ότι πραγματικά θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον μια πολύ επικίνδυνη, σοβαρή κατάσταση, όπου θα πρέπει σίγουρα να μειώσουμε το βαθμό των αντιβιωτικών που χρησιμοποιούμε στον κλάδο της γεωργίας. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να είναι πολύ δύσκολο από τεχνικής ή οικονομικής πλευράς. Πραγματικά θα ήθελα να μπορούσα να είχα συντάξει μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας όπου θα περιέγραφα όλες αυτές τις ανησυχίες που εκφράζουν οι ίδιοι εκτινοτρόφοι, οι οποίοι φοβούνται τελικά ότι το κόστος θα αυξηθεί πάρα πολύ εξαιτίας των εξελίξεων που είχαμε τα τελευταία χρόνια και πολλοί φοβούνται ότι αυτοί θα πληρώσουν το τίμημα όλων αυτών των εξελίξεων που είχαμε στον κλάδο τους τα τελευταία χρόνια. Νομίζω λοιπόν δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τους ανθρώπους αυτούς και τα συμφέροντά τους. Ξέρω ότι ενδεχομένω αυτή τη στιγμή αυτό να το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού, πάντω υποχρέωσή μα, συμμετέχοντα στην Επιτροπή αυτή, να μην ξεχνάμε και του ίδιου του κοινοτρόφου. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Πάλσεν για την ε, για τη δουλειά 15-16 συζήτηση 21 Σεπτεμβρίου Ιουλίου και 21 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή ΕΜΒΗ. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα. τροποποίηση του κανονισμού 726 του 2004 για θέσει κοινοτικών διαδικασιών χορήγηση άδειε και υποπτία όσον αφορά τα φάρμακα που προέρχονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου, Στάνισλαβ Πόλτσακ, ο συντάκτη νομοδότηση. ΕΝΒΙ, Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή. Έχουμε τροπολογίε. Στενή σχέση αυτού του σημείου τη μεσαίταξη με το προηγούμενο. Ουσιαστικά μιλάμε για την άδεια και εποπτεία φάρμακων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πόλτσακ για να σχολιάσει τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. διότι τα περισσότερα ζητήματα έχουν ήδη καλυφθεί από την έκθεση της κυρίας Πάουλσεν. Θα αναφερθώ απλώς σε κάποια τεχνικά ζητήματα. Όπως είπατε και εσείς πάντως το θέμα σχετίζεται άμεσα με τα προηγούμενα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Στο παρελθόν, στις προηγούμενες συνεδριάσεις μου, συζητήσαμε κάποια τμήματα της γνωμοδότησης αυτής Συνεπώς θα ήθελα να επικεντρωθώ τώρα στις ε, τροπολογίες που έχουν υπευληθεί, 39 συνολικά είναι οι τροπολογίες αυτές. Ορισμένες ε, καλύπτονται ήδη από την έκθεση της κυρίας Πάουλσεν και αυτό διευκολύνει κάπως το δικό μου το έργο. Σας ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ για την ε, συμβολή σας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε μία ενιαία θέση για το ζήτημα αυτό. Υπάρχουν ε, κάποια, σαφώς κάποια κίνδυνοι για το περιβάλλον. Βεβαίως είναι και πολύ καλή ιδέα, αλλά κατά κάποιον τρόπο θα πρέπει να μπούμε τα κεντρικά σημεία αυτής της ιδέας και φοβάμαι ότι δεν έχει υπάρξει πολύ καλή έρευνα. Να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες προκύπτουν αυτέ οι μονογραφίες. Ε, η κτηνιατρική βιομηχανία έχει καταθέσει την πρόταση ότι θα πρέπει να δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των μελετών. Οι μελέτες αυτές βεβαίω είναι μια πολύ καλή επιστημονική βάση, αλλά φοβάμαι ότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος ε, έτσι ώστε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα να συμπεριληφθούν στην έκθεσή μου. και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μία ενδελεχέστερη συζήτηση ε, σχετικά με τους κινδύνους αυτών των ουσιών για το περιβάλλον. Κατά την άποψή μου, αυτό που έχει σημασία είναι ποιο είναι το βάρος αυτής της έκθεσης. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ τεχνικό και νομίζω ότι πρέπει να επιδιώξουμε τη συμφωνία ε, σχετικά με τις ε, τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Άλλωστε είπα κάποια πράγματα και για την προηγούμενη έκθεση. Να ευχαριστήσω πάντως τον εισηγητή. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα τεχνικό. Έχουν υποβληθεί κάποιες τροπολογίες για τις οποίες νομίζω θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμβαστική πρόταση. Ήδη έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια αυτή με τον εισηγητή. Με ενδιαφέρει πάντως ιδιαίτερα τα όσα λέει η κυρία Σκορκέιτον το να δημιουργηθεί δηλαδή μια βάση δεδομένων η οποία θα επικαιροποιείται τακτικά προκειμένου να γνωρίσουμε πραγματικά ποιε είναι οι δραστικέ ουσίε των ε, κτηνιατρικών φαρμάκων. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συμπεριλάβουμε την πρόταση αυτή και στην έκθεση αυτή και κυρίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τονίσει ότι είναι αναγκαίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων να διατηρήσει τον υφιστάμενο ρόλο που έχει για την αδειοδότηση των κτηνιατρικών φαρμάκων μέσω της κεντρικής μεθόδου αδειοδότησης και κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα υπάρχει μια καλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στον κανονισμό 726 και στον νέο κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, η ε, κυρία Αγιούζο έχει το λόγο. Ε, θα είμαι πολύ σύντομη κύριε Πρόεδρε. Αυτός ο διαχωρισμός ε, των οργανισμών είναι απολύτως απαραίτητος και θέλω να παραμείνει το ερώτημα. Χρειαζόμαστε αυτούς τους οργανισμούς ή καλύτερα να παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν. Απλά πολλαπλασιάζονται αυτοί οι οργανισμοί στην Ευρώπη και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί χρειαζόμαστε αυτό το νέο οργανισμό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με λύπη βλέπω για μία ακόμη φορά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μία απλοποίηση ενός κείμενου, ενός φυστάμενου κανονισμού, μόνο και μόνο για να επιβάλλει για μία ακόμα φορά αυτό το οποίο ονομάζουμε στα γαλλικά ουζίνα γκάζ, δηλαδή ένα πολύ πολύπλοκο σύστημα. Το κόστος του νέου αυτού Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων βασίζεται εκταρχά σε μία αύξηση των τελών και σε μία αύξηση τη τελική τιμή των φαρμάκων. Και με ιδιαίτερη ακόμα λύπη βλέπουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μολονότι θα έπρεπε να γνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η πρώτη υπεύθυνη για την πληθώρα αυτή των κανονισμών, ανταυτού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται συνένοχο τη περαιτέρω αυτή ε, νομοθετικής προσπάθειας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζαμε ότι θα μπορούσαμε εμπροκειμένου να είχαμε απλουστεύσει πολύ περισσότερο τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σκοτ Κατώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι εδώ έχουμε να προστατεύσουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, να παίξουμε την δημόσια υγεία και την υγεία των ε, ζώων, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην συγχαίουμε τους κανόνες για την προστασία της υγείας με τη γραφειοκρατία και οφείλουμε να διασφαλίσουμε αυτός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων να έχει και τα απαραίτητα κονδύλια. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να μην επιβάλλουμε περιορισμό και περικοπή των κονδυλίων, γιατί αλλιώς ε, θα διαπιστώσουμε μακροπρόθεσμα ότι υπάρχει κρίση στην υγεία των ζώων και στη δημόσια υγεία και αυτό θα μας κοστίσει πολύ περισσότερο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να συσταστεί αυτός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός και να πρικοδοτηθεί και ε, δεόντως. Έχω λοιπόν να θίξω ορισμένα θέματα. Πρώτον, με μεγάλη ανησυχία βλέπω ότι προτείνεται για τον οργανισμό αυτό περιορισμένο προσωπικό. Ε, που θα εφαρμόζει τους κανόνες. Ε, φτάνει αυτό το προσωπικό για να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνεται η απαραίτητη συλλογή δεδομένων, η ανάλυση τους που είναι απαραίτητα για να υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσης, αντιμετώπισης της αντοχής ε, στα αντιβιωτικά, κάτι που είναι μεγάλη απειλή. Ο οργανισμός αυτός παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, η επιστημονική του ε, ε, γνώμη είναι, πολύ, είναι καθοριστική. Επίσης πιστεύω ότι χρειαζόμαστε επαρκείς πόρους για να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που θα αποκτάμε για τα ευρωπαϊκά φάρμακα. Στο σχετικό κανονισμό προβλέπεται ότι αυτός ο οργανισμός θα αναθεωρήσει ε, τις αδειοδοτήσεις. Θεωρούμε ότι πρέπει λοιπόν να έχει τους απαραίτητους πόρους και εν πάση περιπτώσει αν δεν υπάρχουν ε, απαραίτητες ανανεώσεις για τα φάρμακα η φαρμακοεπαγρύπνηση πρέπει να είναι πολύ πιο ισχυρή. Χαίρομαι που ενδιαφέρεται και ο κύριος Καπούτο για την επικαιροποιημένη ε, βάση δεδομένων. Θα συμφωνήσω με μια σχετική τοπολογία και θα συζητήσω με τους ε, υπόλοιπους για, και για άλλες τροπολογίες. Πρόεδρος, ε, λοιπόν, νομίζω ότι συζητήσαμε επαρκώς και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, αλλά πριν από αυτόν άλλος ένας ε, συνάδελφος θέλει το λόγο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Κοιτάξτε, όσον αφορά το μεγάλο θέμα, κατά πόσον χρειαζόμαστε την εξουσιοδότηση, όχι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι περνάνε πολλά καλά ψηφίσματα και καλοί κανονισμοί, εντάξει και κάποιοι κακοί, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε τη ε, δυνατότητα παρακολούθησης. Τι γίνεται στα Εθνικά Κοινοβούλια, είμαι σίγουρος ότι ας πούμε για άλλα θέματα ε, εγκληματικά εκεί υπάρχει αστυνομία και επιβάλλονται και τιμωρίες. Θέλω να υπάρχει ένας οργανισμός που θα εξετάει σωστά τα γεγονότα, τα στατιστικά δεδομένα και να μπορεί και να ενημερώνει την Κομισιόν εφόσον δεν εφαρμόζονται σωστά οι κανονισμοί στα κράτη-μέλη. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι σε όλα τα κράτη-μέλη θα είναι καλή και η ε, παρακολούθηση. Τεχνικό το θέμα, αλλά αν τελικά θέλουμε να πετύχουμε πρέπει ε, τουλάχιστον για κάποια μερική επιτυχία να μεριμνήσουμε ε, για την υγεία των ζώων και ίσως μπορούμε και στο μέλλον να μεριμνήσουμε για ένα απλούστερο κανονισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος, πολύ πιο σύντομος ε, από ό,τι πριν πρώτον. Για ποιο λόγο υποβλήθηκε η πρόταση αυτή σε συνδυασμό με την προηγούμενη πρώτον, διότι πρέπει να τροποποιήσουμε τον κανονισμό 726 του 2004, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τώρα η διαδικασία κεντρική αδειοδότησης να ενσωματωθεί σε έναν νέο κανονισμό μαζί με, τις άλλες, ε, με τους άλλους κανονισμούς αδειοδότησης. Να ισχύει δηλαδή και για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Και θέλουμε ο νέος κανονισμός να συνάδει με τη συνθήκη της Λισαβόνας και τις σχετικές διατάξεις. Αυτό προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε. Δεν θα θέλαμε να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της αναθεώρησης για να συμπεριληφθούν και νέες αρμοδιότητες για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ή για άλλου εμπλεκόμενου φορείς. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις που ακούσαμε σήμερα, πρώτον να πω ότι πρέπει να σας διαβεβαιώσω, να διαβεβαιώσω κυρίως την κυρία Γιούσο και τον κύριο Φεγό, ότι δεν προβλέπεται ένας νέος οργανισμός, αναφερόμαστε πάντα στον υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Δεν υπάρχει λοιπόν κύριε Θεό κάποιο νέο ευρωπαϊκό θεσμό, ο οποίο δημιουργείται αυτή τη στιγμή. Δεν περιπλέκουμε εμεί περισσότερο τα πράγματα. Ξέρετε ότι υπάρχει εδώ και 20 χρόνια αυτό ο οργανισμό, λειτουργεί πολύ καλά. Δεν προτείναμε σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί κάποιο νέο οργανισμό. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Κόπκε και την κυρία Φέντερ, και τον κύριο Φέντερλε ότι όντω θα πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα μέσα τα οποία να συνάδουν με τι φιλοδοξίε μα, θα πρέπει να έχουμε του απαραίτητου πόρου. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει περίπου 800 υπαλλήλους Όσοι ασχολούνται με τα κνητικά φάρμακα δεν είναι πολύ αριθμοί, πάντως σας διαβεβαιώ ότι έχουμε συζητήσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κάθε δυνατή λεπτομέρεια με τους συναδέλφους και τους φίλους που έχουμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και μόνο συνέχεια υποβάλαμε επίσημα την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι δεν δημιουργούμε ένα νέο οργανισμό, δεν περιπλέκουμε τα πράγματα, θέλουμε ουσιαστικά να διευκολύνουμε την ομαλή λειτουργία αυτού του ήδη φυστάμενου Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά την αδειοδότηση και όσον αφορά το σύστημα παρακολούθηση των κτηνιατρικών φαρμάκων. Σα ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ε, ο εισηγητή, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Να πω τελειώνοντας Ελπίζω μαζί με τους ε, σκιώδεις ηγητές θα μπορέσουμε να καταθέσουμε ε, συμβαστικές τροπολογίες. Ε, δεν υπάρχουν τόσες πολλές τροπολογίες και θέλω να πω το εξής στην Κομισιόν. Ο νέος κανονισμός αλλάζει την κατανομή των αρμοδιοτήτων. Η Επιτροπή έχει επεξεργαστεί και τον αντίκτυπο επιπτώσεων και κατά την άποψή μου αυτά ε, δεν ε, είναι υπέρ του οργανισμού. Το λέω κιόλας ε, στη δική μου την εισήγηση. Η πρικοδότηση του οργανισμού θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη χρηματοδότηση του συστήματος και επίσης θα υπάρχουν και επιπτώσεις ε, οικονομικής φύσεως στα κράτη-μέλη. Θα υπάρχουν επιπτώσεις ε, στους προεπλογισμούς των κρατών μελών. Γι' αυτό, κατά την άποψή μου, θα πρέπει οι αρμοδιότητες ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατανεμηθούν διαφορετικά. Ο κύριος Φεράων πρέπει να συμφωνήσει Όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε κατά νου και να δεχτούμε ότι πρέπει να κατανοηθούν διαφορετικά οι αρμοδιότητες. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στις 15 και 16 Ιουλίου ε, θα συζητηθεί, θα ψηφιστεί η έκθεση αυτή. Στις 22 Σεπτεμβρίου θα συζητηθεί στην Επιτροπή ΕΝΒΗ και τώρα πάμε στο 8ο σημείο της ημερήσιας διάταξης, η δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Άλμπερτ Dess και ε, καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι Επιτροπή Περιβάλλοντος. Komisji Λοιπόν, η δική μας Επιτροπή έχει δεσμευτεί να γνωμοδοτήσει κυρίως όσον αφορά στη δυνατότητα των κρατών μελών να χρησιμοποιούν ε, γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωτροφές στην επικράτειά τους. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πριν από τη Σε σχέση αυτού του θέματος δεν υπήρξε πλειοψηφία υπέρ αλλά ούτε και κατά. Και έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την απόφαση με βάση την νομοθεσία που ισχύει σήμερα αλλά χωρίς ε, να υπερψηφιστεί το θέμα στην Επιτροπή. Ο κανονισμός 1829 του 2003 επιτρέπει στα κράτη-μέλη να προβαίνουν σε περιορισμούς ή απαγόρευση ως προς την χρήση των ε, γενετικώς ε, τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών, αλλά αυτό βέβαια μόνο εφόσον τα κράτη-μέλη είναι σε θέση να αποδείξουν ότι αυτοί οι οργανισμοί αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον ή για την υγεία. Η αξιολόγηση ποικίλει, πολλές και διαφορετικές αξιολογήσεις Εδώ λοιπόν θα συζητήσουμε για την αναθεώρηση αυτού του κανονισμού και για τη δυνατότητα να οριστεί ένα πλαίσιο έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν στην επικράτειά τους να λάβουν μέτρα τα οποία ε, θα αποσκοπούν να απαγορεύονται ή να περίζονται οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί Αυτή λοιπόν η γνωμοδότηση έχει αποδοθεί στον κύριο Ντές. Αλλά πριν λάβει το λόγο ο κύριος Ντές, καλύτερα να λάβει το λόγο η Κομισιόν για να μας εξηγήσει ποιος είναι ο στόχος αυτής της ε, πρωτοβουλίας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, honorable members. Σας ευχαριστώ πολύ, αξιότιμοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω εν συντομία την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροπή του κανονισμού περί τροφίμων και ζωοτροφών. Γνωρίζετε ότι το λόγο σχέδιο νομοθετικής πρότασης απορρέει από τη δέσμη κατευθυντήμων γραμμών που ενέκρινε τον Ιούλιο του 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόταση πρέπει να ειδωθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και συγκεκριμένα με βάση το γεγονό ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες σε πολλά κράτη-μέλη είναι επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά τους ε, γενικούς τροποποιημένους οργανισμούς. Ταυτόχρονα όμως πολλοί παραγωγοί εξαρτώνται από εισαγωγές 32 εκατομμύρια τόνου σόγια στο χρόνο εισάγουμε και στι περισσότερε περιπτώσει πρόκειται για μεταλλαγμένη σόγια. Παράγουμε μόλι 1,4 εκατομμύρια τόνου. Δείτε την αναλογία. Λιγότερο δηλαδή του 5% των αναγκών που έχουμε. Αν δηλαδή θέλουμε να αυξήσουμε την παραγωγή, να καλύπτονται οι ανάγκες μας, σημαίνει ότι η παραγωγή πρέπει να αυξηθεί 20 φορές. Φυσικά ανεδαφικό κάτι τέτοιο. Λόγω του διλήμματος ε, υπήρξε πόλωση της χρήσης όταν χρειάστηκε να ψηφίσουν υπέρ κατά της χρήσης των κατά την εύσα ασφαλος ασφαλών μεταλλαγμένων. Από τα 67 λοιπόν τέτοια προϊόντα έχουμε ε, ειδική πλειοψηφία υπέρ Μάλλον δεν υπήρξε ειδική πλειοψηφία υπέρ ούτε κατά. Of the time. The Commission has therefore always taken alone the Αφού στο Συμβούλιο λοιπόν δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που μετά από μελέτη αντικτύπου προσπαθεί να εφαρμόσει τις νομικές της υποχρεώσεις, γιατί είναι νομική υποχρέωση του Κομισιόν, για αυτά τα τρόφιμα, τα μεταλλαγμένα. Μια μοναδική κατάσταση στην ιστορία της επιτροπολογίας. Αυτό οδήγησε σε ένα δημοκρατικό έλλειμμα για το σύστημα, όπως τουλάχιστον δεν λαμβανόμαστε και αυτό είναι σε βάρος όλων. Καλούμε λοιπόν όλους αυτή τη στιγμή να λάβουν τις ευθύνες τους. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πλέον ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε το status quo και θεωρούμε επίσης ότι οι συζητήσεις από τις προτάσεις αυτής είναι πολύ σημαντικές και θα βοηθήσουν να διευκρινιστεί η κατάσταση, να ξεκαθαρίσει το θέμα και να εξευρεθούν οι απαραίτητε λύσεις και να ληφθούν οι απαραίτητε αποφάσει. Η αναθεώρηση τη διαδικασία λήψη αποφάσεων για την ε, αδειοδότηση μεταλλαγμένων κατέληξε στο ότι η καλύτερη λύση είναι να επεκταθούν οι διατάξεις της νέας Οδηγία που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο για την καλλιέργεια μεταλλαγμένων και στα γενετικώ τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές σήμερα βλέπουμε να υπάρχουν σημαντικέ αδυναμίε και ελλείψει. Πρώτον, η αλλαγή του κανονισμού επιτροπολισμών για του μεταλλαγμένου οργανισμού θα οδηγούσε σε διακρίσει. Γιατί να αλλάξουν οι κανόνε μόνο για μεταλλαγμένα Πώς απαντάει κανείς αυτό το ερώτημα. Επίσης, η αλλαγή των ε, κανόνων ε, ψηφοφορίας. Πώς θα αλλάξει αυτό αφού κατοχυρώνονται στη συνθήκη για να υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση των 28 κρατών μελών. Άρα αλλαγή θα σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε και τη συνθήκη. Τέλος, το να δώσουμε ξανά πίσω στα κρατημέλη τα αρμοδία όταν αποφασίζουν για αυτές τις εγκρίσεις των μεταλλαγμένων δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει γιατί σημαίνει ότι θα δεχόμασταν και διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας μεταξύ των κρατών μελών. Άρα, στην ουσία η πρόταση της Κομισιόν θα δώσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να λάβουν υπόψη τις εθνικές συνθήκες, να περιορίζουν να απαγορεύουν τη χρήση εξουσιοδοτημένων, μάλλον εγκεκριμένων γενικοστοπευμένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους. Έτσι θα έχουμε περισσότερη επικουρικότητα στο σύστημα, ώστε η τελική επιλογή να είναι πλέον πιο κοντά στους εθνικούς ε, υπηκούς πολίτες των κρατών μελών. Γιατί τώρα μπορεί κάποιο κράτο για άλλου λόγου και όχι για ησυχία ασφάλεια να απέχει από την ψηφοφορία. Δεν αλλάζει με την πρόταση όμω η χορήγηση των αδειών στου γενετικους τροποποιημενου προκειμένου. Επίση, αποφάσεις opt-out θα πρέπει να είναι συμβατέ με τις βασικέ αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή οι πολίτε πρέπει να μπορούν να απολάβουν ενό επίπεδου προστασία, Δηλαδή η αξιολόγηση του αντικτύπου και η αξιολόγηση των ε, γενικών στροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών θα πρέπει να γίνεται με ομογενή τρόπο και θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί, ε, σοβαστές, σεβαστές αντικτύπου και εκτίμηση κινδύνου της ΕΦΣΑ. Έχουμε και τον κανονισμό της ρήτας διασφάλισης. Ισχύει. Δεύτερον, τα μέτρα opt-out θα πρέπει να συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και τους κανόνες της ιστορικής αγοράς. Τέτοιες αποφάσεις λοιπόν θα πρέπει πρώτα να βασίζονται σε προεξάρχοντες ε, λόγους για εθνική υγεία και να είναι αναλογική και μη διακριτική. Τα κράτη-μέλη μπορούν να απαγορεύσουν μόνο τη χρήση γενετικώ τροποποιημένο τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά του. Δεν μπορούν να απαγορεύσουν την ελεύθερη κυκλοφορία τη εισαγωγή. Άμα αποφασίσουν λοιπόν να περιορίσουν, να απαγορεύσουν τη χρήση μεταλλαγμένων τροφίμων και ζωοτροφών, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξετάζουν πολύ προσεκτικά τον κοινωνικό, οικονομικό αντίκτυπο των αποφάσεων του για την αλυσίδα και τη διάδοση με τι ε, πώληση τέτοιων τροφίμων και ζωοτροφών. οι πολίτες και οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις θα έχουν περισσότερο λόγο. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε κάποια ζητήματα. Υπάρχουν πολιτικές προκλήσεις και αυτές μπορούν να λυθούν ιδίως σε μια εποχή που έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Σας ζητώ λοιπόν ο όλους κύριε Πρόεδρε, κύριε Σεγητά, αγαπητοί βουλευτές, να ξεκινήσετε επικοδομητικό διάλογο για να προχωρήσουμε με την νομοθετική διαδικασία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Λοιπόν, ε, είχα ακούσαμε την Επιτροπή. Τώρα, ε, δίνω το λόγο στον κύριο Ντές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα αφήσω την ε, εισαγωγή κατά μέρο γιατί εσεί ω ε, πρόεδρο και η Επιτροπή παρουσιάσετε με τον κανονισμό 1829 του 3 ε, πλέον υπάρχει αυταρρυσία στην αγορά. Οι εθνικές απαγορεύσει δεν συμβαδίζουν με το διεθνές δίκαιο, οδηγούν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού αν δεν στηρίζονται από σοβαρέ επιφυλάξει για την υγεία την πρόταση της Επιτροπής δεν θεωρώ ότι πρέπει να τη στηρίξουμε. Δεν μας βοηθάει στο να επιτύχουμε το στόχο μας. την πρόταση αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να αποδείξουν το κατά πόσον τα δικά τους ε, τα μέτρα συμβαδίζουν με τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγορά, ε, για τις διεθνείς υποχρεώσεις και για τον ΠΟΕ. Με αυτή την πρόταση, κατά την άποψή μου, η εσωτερική αγορά Πρέπει άραγε να εισάγουμε και πάλι εμπορευματικούς φραγμούς ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη. Ποιο είναι το επίπεδο ανοχής. Υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την εισαγωγή προϊόντων. Ο κύριος Γιούγκερ είπε ότι θέλει να περιορίσει τη γραφειοκρατία. Εδώ όμως δημιουργείται ένα τέρας της γραφειοκρατίας. Οι Υπουργοί Γεωργίας όλων των πολιτικών τάσεων είπαν ότι θα πρέπει να αναπεμφθεί αυτή η πρόταση. Εδώ υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Αυτό το τέρας γραφειοκρατίας πρέπει να αναπεμφθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η Επιτροπή φέρει μεγάλη ευθύνη ε, σε αυτό το πλέγμα των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα αφήσουμε όλο αυτό το θέμα στην Επιτροπή. Και η απόφαση της Επιτροπής δεν είναι συνεπής και με άλλες ε, ε, αποφάσεις. Ο κ. Τσόλος το 7% της παραγωγής να αφαιρεθεί και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο κατόρθωσε σε αυτές τις εκτάσεις ε, να καλλιεργούνται άλλα ε, προϊόντα όπως μπιζέλια, Πασόλια, ε, Μπορούμε λοιπόν σε αυτές ε, τις εκτάσεις να καλλιεργούμε όσπρια και δεν χρειαζόμαστε ή χρειαζόμαστε λιγότερες εισαγωγές. Εδώ λοιπόν η Κομισιόν έκανε τελείως λανθασμένη τελειως έλαντασμένη όπως συνέβη και με τη γεωργική μεταρρύθμιση. Επίσης ε, μίλησα και με εκπροσώπους Επιτροπής ΕΝΒΗ. Δεν θέλω να προκαταλάβω τίποτα αλλά θέλω να σας πω ότι κατά την άποψή μου στην ΕΝΒΗ διαφαίνεται μεγάλη πλειοψηφία στο να αναπεμφθεί αυτή η έκθεση. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η έκθεση γιατί σε τελική ανάλυση αντιβαίνει στην ελευθερία της αγοράς μας. Και γι' αυτό προτείνω εμείς στη γνωμοδότησή μας ε, να ακολουθήσουμε την ίδια θέση όπως και η και να αναπέμψουμε την έκθεση αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή σας την ε, άποψη, την παρουσίαση της άποψής σας. Ξεκινάει λοιπόν η συζήτηση. Έχουν ζητήσει το λόγο πάρα πολλοί συνάδελφοι. Στις 6.30 ξεκινάνε δύο άλλες σημαντικές συναντήσεις η συνάντηση του κυρίου Νίκολσον για την ανταγωνιστικότητα του τομέα των αυγών. Θα συζητηθεί επίσης το TTP. Ο κύριος ε, Νίκολσον, εκείνος που έχει οργανώσει αυτή τη συνάντηση και η Κόπα Κοσέκα και αυτοί στις 6.30 έχουν συνάντηση κάτω στο σαλόνι. Εκεί θα μιλήσουν για το γάλα, για την κατάσταση στο γαλακτοκομικό τομέα. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να συμμετάσχουμε και στις δύο αυτές ε, εκδηλώσεις γιατί όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά και θα ήταν καλό να πάμε και στις δύο εκδηλώσεις. Λοιπόν, για 1,5 λεπτό ο καθένας, όχι παραπάνω. Νομίζω ότι το θέμα είναι γνωστό, ε, μπορούμε να πούμε πολλά, αλλά και πολύ λίγα. Εγώ λέω να πείτε λίγα. Ο κύριος Μποβάν. έχει το λόγο. Euh, Πρόεδρε, κοιτάξτε, ε, για μία φορά συμφωνώ με τον κύριο Ντέσε. Επί της ουσίας το κείμενο αυτό δεν είναι καλό. Έχει πολύ κακή δομή, κακή διάρθρωση, όπως και το πρώτο κείμενο που είχαμε για τις καλλιέργειες. Και έχουμε ουσιαστικά εδώ πέρα το ίδιο κείμενο. Μας προκαλεί εντύπωση το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν το κείμενο για τους σπόρους και θα απορρίψουμε τελικά το κείμενο που έχει να κάνει με τα τρόφιμα. Δεν πειράζει, τόσο το καλύτερο. Ας δημιουργηθεί και λίγο αναστάτωση. Βλέπετε ότι η προτινόμενη νομοθεσία είναι κακή, είναι ήδη κακή νομοθεσία και για τους σπόρους βέβαια. Σήμερα η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται εδώ πέρα και αναγνωρίζει και δεν θα δώσω ονόματα. Πάντως ανταλλαγές που είχαμε εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν είναι δυνατόν να περασπιστεί τη θέση της ενώπιον του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Δηλαδή δεν μπορούμε να βασιστούμε στον κανονισμό SPS προκειμένου να υπερασπιστούμε τα κράτη μας αν δεχθούμε επίθεση ή αν γίνει προσφυγή από κάποιο άλλο κράτος του ΠΟΕ. Και μπορούμε να βασιστούμε τελικά για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς μόνο στους, μη, μόνο στα, στο μέσο των μη δεσμολογικών εμποδίων. Ξέρετε όμως ότι δεν μπορούμε να δώσουμε μάχη χρησιμοποιώντας μόνο αυτό το μέσο. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι καλό το κείμενο αυτό και ότι δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Που έγκυται τώρα το πρόβλημα. Το πρόβλημα έγκυται στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα αρνείται μολυνότι το ζητά ο κύριος Γιούγκερ να εξετάσει εκ νέου το σύνολο των νομοθετημάτων που έχουν να κάνουν με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς όσον αφορά την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνικο-οικονομική πτυχή όλων αυτών των νομοθετημάτων. Αν δεν εξετάσουμε την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική πτυχή των νομοθετημάτων αυτών θα καταλήξουμε σε ένα σαθρό νομοθέτημα το οποίο δεν θα μπορέσουμε ποτέ να υποστηρίξουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή μας ζητά απλώς να λυγίσουμε μπροστά στις μεγάλες αυτές επιχειρήσεις, τις πολυεθνικές, οι οποίες επιβάλλουν και υποστηρίζουν τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Είναι οι επιχειρήσεις αυτές οι οποίες θέλουν να διευκολύνουν την πρόσβαση των δικών τους προϊόντων στο έδαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε, αν έχει την καλοσύνη, μην επαλαμβάνετε αυτά που έχουν λεχτεί Η κυρία Μπετία. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και κύριε Ντέ, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Καλωσορίζουμε τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορούν να αποφασίζουν για την χρησιμοποίηση των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να καθορίσουμε ξεκάθαρα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευση της χρήσης γενικών τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικρατεία στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού προβλέπει τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν να απαγορεύουν τη χρήση μεταλλαγμένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους. Να επιστήσω επίση την προσοχή σας στο γεγονός ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε την ε, το πώς τα κράτη-μέλη μπορούν να περιορίζουν ή να απαγορεύουν αυτή τη χρήση των μεταλλαγμένων τροφίμων και ζωοτροφών και πώς αυτό συνάδει με τις διεθνείς συμφωνίες εμπορίου που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη θα μπορούν κατά την άποψή μου να αποφασίζουν τον περιορισμό Η την απαγόρευση χρήσης μεταλλαγμένων τροφίμων και ζωοτροφών χωρίς να αιτιολογούν την απόφαση αυτή. Η πρόταση του κανονισμού επίσης θα πρέπει να ρυθμίζει στους λόγους που θα μπορούσαν να επικαλεστούν λογικά τα κράτη-μέλη για τον περιορισμό της απαγόρευση της χρήσης μεταλλαγμένων τροφίμων και ζωοτροφών προκειμένου να προασπίσουν τα εθνικά τους συμφέροντα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς που ήσασταν σύντομος, η κυρία Χόλμπους. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, νομίζω σήμερα το θέμα δεν είναι το να επιτρέψουμε ειδικέ άδειες στην Ευρώπη για τα γενετικά μεταλλαγμένα. Το θέμα είναι με βάση κάποια κριτήρια θα επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτών των τροφίμων και των ζωοτροφών που είναι γενετικά μεταλλαγμένα. Κοινωνικο-οικονομική, πολιτική, άλλοι λόγοι παίζουν σαφώς ρόλο, τα αναφέρατε σήμερα. Αλλά θέλω να επισημάνω το εξής, η ΕΦΣΑ έχει τις επιστημονικά τεκμηριωμένες αντιρρήσεις των κρατών μελών για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Έτσι λοιπόν, τι συμβαίνει ο αραβόσιτος και άλλες διασταυρώσεις από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, όλα αυτά εμφανίζονται στην αγορά και παρουσιάζονται ως τρόφιμα που δεν συνεπάγονται κανένα κίνδυνο. Αυτά όμως δεν έχουν δοκιμαστεί ούτε σε μελέτες ούτε πουθενά αλλού. Υπάρχουν επιστημονικές αντιρρήσεις, δυστυχώς όμως αυτές ε, μπαίνουν κάτω από το τραπέζι και τώρα καταβάλλεται προσπάθεια όλο αυτό να ε, μεταφερθεί στους ώμους των ε, κρατών μελών. Ο κύριος Γιούγκερ ήθελε να καταργήσει κύριε Ντες, όχι μόνο τη γραφειοκρατία αλλά στην αρχή είχε πει ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης της ΕΦΣΑ είναι μη επιστημονικές και αντιδημοκρατικές. Αυτά είναι τα λόγια του και πρέπει πάνω σε αυτά να βασιστούμε. Χρειαζόμαστε επιστημονικά τεκμηριωμένα κριτήρια, πάνω σε αυτά θα πρέπει να βασίζονται οι αντιδιωτήσεις και αν τηρούνται όλα αυτά τότε να κυκλοφορούν τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Πρέπει να πω στην Επιτροπή σας ότι εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο Ζωζέ Μποβέ, ο οποίος στο παρελθόν έχει καταστρέψει τέτοιες καλλιέργειες γενετικώς τροπημένων τροφίμων, συνομιλεί εδώ πέρα με μένα τον ίδιο, ο οποίος έχω καλλιεργήσει τέτοια τρόφιμα. Δεν μιλάμε όμως εδώ πέρα για την καλλιέργεια, μιλάμε για την χρήση των τροφίμων αυτών και των ζωοτροφών αυτών και 32 εκατομμύρια τόνοι εισάγονται, μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα τους υποκαταστήσουμε αυτούς. Εγώ ασχολούμαι με τον τομέα των αυγών ελευθέρας βοσκής στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν χρησιμοποιούμε γενικά τροποποιημένες πρωτεΐνες, αλλά είναι πολύ δύσκολο να καταφέρνουμε να εισάγουμε καθαρούς σπόρους σόγιας ακριβώς επειδή δεν μπορούμε τελικά να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη ιχνηλασιμότητα. Χρειάστηκε εγώ να πληρώσω επίσης 680 λίρες ανατόνο για μη τροποποιημένη σόγια από το Καζακστάν και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Θα πρέπει ουσιαστικά να σκοτώσω τα πτηνά μου γιατί δεν είμαι σε θέση να τα θρέψω σωστά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε το ζήτημα αυτό. Οι πωλήσει από την άλλη δεν επηρεάζονται καθόλου από το αν τελικά έχει θρέψει κανείς τα ζώα του με γενετικά τροπημένους οργανισμούς ή όχι. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι να απαγορεύσετε την εισαγωγή των μεταλλαγμένων αυτών τροφίμων δεν θα καταφέρετε καν να θρέψετε το ζωικό σας κεφάλαιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλλιεργεί κανείς σε μεγάλη κλίμακα μη γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για τη διατροφή των ζώων. Πραγματικά νομίζω ότι περιπλέκει κανείς πάρα πολύ τα πράγματα όταν εμένει σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριο Λουαζό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή δεν μπορούν να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη, έπρεπε να αποφασίσει για αυτά. Περίεργο όμως βασίζεστε στην ε, αμφιβολία για το κατά πόσο είναι ασφαλή αυτά τα τρόφιμα, αλλά ε, έχετε τότε να τα ε, επιτρέψετε και αποφασίσετε για όνομα των κρατών μελολέτε δεν θα υπάρξει κάποια επίπτωση για την άδεια κυκλοφορία των μεταλλαγμένων τροφίμων και ζωοτροφών που ορίζονται σε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό. Υπάρχει και το άρθρο 34 για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Δεν πρέπει να παραβιαστεί διατάξεις αυτών των, αυτού του άρθρου. Τώρα, αν ένα κράτος αρνηθεί τη χρήση αυτών των τροφίμων ζωοτροφών και το διπλανό κράτος τη δεχθεί με την ελεύθερη κυκλοφορία, αποτέλεσμα είναι να έρθουν στη στερική αγορά αυτού του κράτους που δεν τα θέλει αυτά τα τρόφιμα. Απ' την άλλη, σε ό,τι αφορά ε, τη χρήση μεταλλαγμένων τροφών και ζωοτροφών. Η μόνη πολιτική που θα δεχόμασταν εμείς για τα μεταλλαγμένα έχει τρία σημεία. Εθνική έρευνα, εθνική παρασκευή και εθνική κατανάλωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. κύριος Αντρία, καταρχά να πω στην Κομισιόν ότι αν κάνει την πρότασή τη ε, για να σεβαστεί τη δημοκρατική Βουλή και τη διαφάνεια, εμεί εγκρίναμε τη δεκαετία του 92.000 ε, ουσιαστικά την απορρίθμιση και πρέπει να το ξαναδούμε γιατί περισσότεροι πολίτες ε, είναι αντίθετη είτε στην καλλιέργεια είτε στη χρήση μεταλλαγμένων στη τροφική αλυσίδα. Η πρότασή σας δεν μπορεί να εφαρμοστεί διότι τα κράτη-μέλη δεν θα μπορέσουν από νομικής πλευράς να αιτιολογήσουν την επιλογή τους να περιορίσουν να παραγορεύσουν ε, τα μεταλλαγμένα. Ή τέλο πάντων ε, εύκολα μπορεί να προσφύγει κανεί σε, σε βάρο του ε, στο δικαστήριο. Δεν καταλαβαίνω πώ η πρόταση τη Κομισιόν αν εφαρμοστεί δεν θα θέσει υποφυσβήτηση την αρχή τη ενότητα τη ενιαία αγορά και θα έχουμε και πρόβλημα σε εμπορικέ μα σχέσει με το εξωτερικό. Πριν από κάποιου μήνε ε, δώσαμε στα κράτη-μέλη την ελευθερία να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια μεταλλαγμένων στην επικράτειά του. Δεν θα έπρεπε ε, να ε, έχετε υπόψη σας ότι θα δημιουργηθεί εμπορική και νομική διαμάχη με την πρότασή σα γιατί έρχεται σε αντίθεση αυτό που προτείνετε τώρα με αυτό που έχουμε κρίνει για την καλλιέργεια. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că se cam vede care să fie soarta Ευχαριστώ πολύ. Γιατί βλέπουμε που θα καταλήξει αυτή η πρόταση. Τέλο πάντων, το πρόβλημα είναι αλλού και πρέπει να το λύσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ συζητούμε για το τι μπορούν ή δεν μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη, να καλλιεργήσουν, να μην καλλιεργήσουν, να περιορίσουν, να μην απα... να απαγορεύσουν τη χρήση μεταλλαγμών κτλ. Όσο υπάρχουν εισαγωγέ, πάντοτε όμω θα υπάρχει ανισότητα, άνηση μεταχείριση απέναντι στους Ευρωπαίους κτηνοτρόφους. Αν αποφασίσουμε ότι αυτά τα μεταλλαγμένα προϊόντα είναι επιβλαβή για τους πολίτες, για την δημόσια υγεία, για ένα μεγάλο μέρος πολιτών, αν όχι για όλους τέλος πάντων, τότε πρέπει να απαγορευτούν και οι εισαγωγές πολύ απλά. Διότι προσφέρουμε πλεονέκτημα σε επιχειρήσει από την Αργεντινή, δεν ξέρω εγώ από πού αλλού, που μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι δικοί μα στενοτρόφοι δεν μπορούν οι ε, γεωργοί να καλλιεργούν τέτοια προϊόντα. Είτε λοιπόν εγκρίνουμε τα προϊόντα αυτά, είτε τα απαγορεύουμε. Όχι όμω την καλλιέργεια να απαγορεύσουμε μόνο, αλλά και την εισαγωγή του. Έτσι μόνο θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Η άλλη επιλογή ή οποιαδήποτε άλλη επιλογή δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Και για μας και για όλα τα κράτη με τα οποία έχουμε σχέση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, κυρία Νόχιλ παρακαλώ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχει ένα βασικό λάθος που είναι η ΕΦΣΑ. Η ΕΦΣΑ καταλήγει σε μία θέση η οποία κατά την άποψή μου δεν εξυπηρετεί την όλη υπόθεση. Αυτό αναφέρθηκε και από την προαλήζασα και θέλω να το επισημάνω. Η ΕΦΣΑ επιστημονικά δεν είναι σε θέση να τοποθετηθεί και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε και πάρα πολλοί άλλοι η ΕΦΣΑ λοιπόν δεν είναι σε θέση να κάνει την αξιολόγηση. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, με κάθε ειλικρίνεια. Η ΕΦΣΑ είναι πολύ κοντά στη βιομηχανία. Έχει σχέσεις με τη βιομηχανία. Άρα δηλαδή όλες οι προτάσεις που τις κατατέθηκαν εγκρίθηκαν από την ΕΦΣΑ. Εδώ δεν έχουμε δυνατότητα ενός οργανισμού που να φιλτράρει, που να διαφυλάσει τα συμφέροντα της Ευρώπης. Ως εκ τούτου εγώ αμφισβητώ και τις αρμοδιότητες και την ανεξαρτησία της ΕΦΣΑ και ο τρόπος ε, με τον οποίο εξαναγκάζει τα κράτη-μέλη να έχουν καλούς δικηγόρους για να παρεμποδίσουν το ενδεχόμενο των εισαγωγών, αυτό απλά εξυπηρετεί τους νομοματείς που θα κερδίσουν πολλά χρήματα με όλη αυτή την υπόθεση. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να το σκεφτείτε σοβαρά και να αλλάξετε στάση. Πρόεδρος, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε λέει η κυρία Μελιόρ, όσον αφορά ε, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ε, Μπορώ να καταλάβω ότι τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν μόνα τους γιατί τα προϊόντα αυτά έχουν σχέση με το έδαφος. Τώρα όμως μιλάμε για τη μεταφορά, ε, την αποθήκευση των ζωοτροφών και γίνεται και για λόγους για τη χρήση τους όπου μπορεί να υπάρχει opting out. Εγώ Όλα αυτά δεν τα θεωρώ εφαρμόσιμα, αντιβαίνουν στο πνεύμα της κοινή αγοράς και δεν μπορώ να φανταστώ ότι δήθεν με κάποιες ε, τροπολογίες θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτόν τον κανονισμό. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ντες ότι πράγματι εδώ πρέπει να λάβουμε θέση και ο Μουτζούρης τον οποίο μας τον δίνει και μας τον σπρώχνει τώρα η Κομισιόν, να τους τον ξαναδώσουμε γιατί μην ξεχνάμε είμαστε σε συμπληγάδες. Αφενός πρέπει να ικανοποιήσουμε ε, τις ε, επιθυμίες των καταναλωτών και αφετέρου να επιτρέψουμε μια εύρυθμα λειτουργούσα γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Ε, το πρώτο είναι το εξής. Όσον αφορά τους ε, σπόρους, εντάξει αυτοί έχουν σχέση με το δαφός. Έχουμε ήδη καταστρέψει εκεί ε, την κοινή αγορά και τώρα θέλουμε όλα αυτά να τα επεκτείνουμε και στις ζωοτροφές. Θέλω να πω στους αδέλφους, ό,τι και αν πιστεύουν για αυτή τη νέα τεχνολογία, η πρόταση δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Εγώ ζω στα σύνορα με την Τσεχία. Πώς θα ελέγχονται οι μεταφορές των ζωοτροφών, θα πρέπει να εισαχθούν εκ νέου συνοριακοί έλεγχοι. Ε, δεν μπορούμε να ελέγχουμε ζωοτροφές στα σύνορα, ακόμα και μέσα στη Γερμανία. Ε, αν θέλετε να υπάρχει πραγματικό έλεγχος, ε, θα πρέπει να επανέλθουν έλεγχοι ακόμα και ανάμεσα στα κρατήρια. Αυτά δεν γίνονται, άρα απορρίπτεται η πρόταση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι εδώ υπάρχει μία προϊστορία. Υπήρξε συμφωνία, επιστημονική αξιολόγηση και μετά από αυτήν η Κομισιόν και το Συμβούλιο ε, κατέληξαν σε κοινή απόφαση. Οι μεν λένε ότι φταίει η ΕΦΣΑ, οι άλλοι λένε ότι δεν έχει σωστή δομή, ούτε είναι η κατάλληλη. Όμως να σε επισημάνω ότι έχουμε κοινή ευθύνη και οι τρεις θεσμοί να επιληφθούμε του θέματος και να καταλήξουμε κάπου γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Γυρίζουμε γύρω-γύρω από την ουρά μας, ε, στέλνουμε προτάσεις στην Κομισιόν, ε, υποτίθεται για να βρεθεί κάποια λύση. Άρα δηλαδή αναπομπή κύριε Πρόεδρε, αλλά να μιλήσουμε με την ησυχία μας για την ΕΨΑ, για την επιστημοσύνη της. Ε, νομίζω ότι αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Νίκολσον έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ξέρω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά την αδειοδότηση των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και συμφωνώ με την Επιτροπή. Όταν ε, ε, υπόθηκε τουλάχιστον σε μια συνεδρίαση κοινοβουλευτική Επιτροπής την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν είναι βιώσιμο το φυστάμενο καθεστώ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είναι σωστή λύση που προβλέπεται. Το να δίνεται αυτή η δυνατότητα που βλέπετε εδώ πέρα στα κράτη-μέλη, νομίζω ότι θα έχει πραγματικά επιζήμιες επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά και θα επηρεάσει προφανώς και τις εμπορικές μας σχέσεις με τρίτες χώρες στο γεωργικό τομέα. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι η Επιτροπή μας και γενικότερα βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται και εξαρτάται πάρα πολύ από τους γεντικά τροποποιημένους οργανισμούς. 32 εκατομμύρια τόνοι ακούσαμε. Επομένως, το να απαγορεύσουμε τους μεταλλαγμένους αυτούς οργανισμούς σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς να τους παράγουμε τη δική μας, στη δική μας την επικράτεια, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να έχουμε μια νομοθεσία η οποία δεν θα επηρεάζει τη δυνατότητά μας να παράγουμε τρόφιμα. Βλέπουμε όμως ότι παράγω, παράλληλα αυξάνεται ο πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις νέες δημογραφικές τάσει. Έχουμε και επιστημονικά δεδομένα. Δυστυχώς όμως σχετικά με την πρόταση αυτή δεν έγινε η μελέτη αντικτύπου και επίσης ε, υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη που θα χρησιμοποιήσουν opt-out για το οποίο όμω δεν απαιτείται επιστημονική αιτιολόγηση. Πρέπει να δούμε επίση πώ η πρόταση αυτή θα επηρεάσει τι εξαγωγέ των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να αποσύρει την πρόταση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρώ ότι και η Επιτροπή Περιβάλλοντο αυτό ακριβώ θα ψηφίσει. Θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή τη, καθότι πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει ω έχει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αγιούσο. Έχουμε ένα πρόβλημα πραγματικά διότι εξαρτώμεθα αλλά και θα συνεχίσουμε να εξαρτώμαστε ιδίω ε, για να θρέψουμε τις, ε, τα ζώα, το ζωικό κεφάλαιο, θα εξαρτώμαστε λοιπόν από τα μεταλλαγμένα προϊόντα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι η ΕΦΣΑ δεν είναι αρμόδια ή δεν είναι αυστηρή. Το Δεκτικό Συμβούλιο της ΕΦΣΑ δεν παρεμβαίνει στην επιλογή των επιστημόνων. Οι επιστήμονε των διαφόρων επιτροπών, των διαφόρων πάνελ, ε, είναι αυθεντίε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είχα την ε, δυνατότητα να είμαι παρατηρητή στην εκλογή των ε, επιστημονικών αυτών συνεργατών. Είδα τα βιογραφικά του σημειώματα. Είναι ικανότατα με υψηλό επιστημονικό επίπεδο άτομα και φυσικά γνωμοδοτούν και έπειτα ε, αναλύονται αυτές από άλλους εμπειρογνώμονες. Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων, διότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν επηρεάζει τις γνωμοδοτήσεις της ΕΦΣΑ, τις οποίες καταρτίζουν απόλυτα ικανοί εμπειρογνώμονες, επεπειραμένοι, με προσόντα. Είχα τη δυνατότητα, όπως είπα, να είμαι της σε ε, τέτοιες ε, διαδικασίε εκλογή μελών πάνελ. Τώρα, αν δεν μα αρέσουν οι γνωμοδοτήσει τη ΕΣΑ, δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίνει οι επιστήμονε που τη συνέταξαν. Πρόκειται για πάρα πολύ αυστηρούς ε, εμπειρονόμες αυστηρές εκθέσεις. Χρησιμοποιούμε αυτούς τους ε, μεταλλαγμένους. Δεν θέλουμε να τους καλλιεργούμε, να μην τους καλλιεργήσουμε, αλλά να πούμε τώρα ότι θα υποκαταστήσουμε ε, με πιζέλια τη φασόλια, τη σόγια, ε, μπορεί τα μένα είναι πράσινα και μακρόστενα και τα άλλα να είναι πράσινα και στρογγυλά, αλλά το θέμα είναι πώς θα θρέψουμε τα ζώα. Everything at this stage has been said. Σε Στη φάση αυτή υπόθηκαν τα πάντα. Δεν υπάρχει λόγος να επαναλάβω τα όσα είπαν οι προαλήσεις. Σας Ευχαριστώ. Piękne wystąpienie, bardzo dziękuję. Pani poseł Kadenbach. Jetzt muss ich widersprechen. Κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω ότι ελέγχθησαν τα πάντα. Ας πούμε, δεν επισημάνθηκε ακόμα το τι περίεργαν όλα αυτά που γίνονται στο Κοινοβούλιο. Εγώ είμαι μέλος Επιτροπής ΕΝΒΗ και μέλος Επιτροπής Άγκρη και πρέπει να σας πω ε, δεν έχω ζήσει ποτέ να συμφωνούμε όλοι και η Επιτροπή Γεωργίας και η Επιτροπή Περιβάλλοντος και οι μεμονωμένες πολιτικές ομάδες ε, να συμφωνούμε όλοι ε, για ένα θέμα. Νομίζω σήμερα συνέβησαν πάρα πολλά εκφράστηκαν πάρα πολλές επιφυλάξεις. Ο πρόεδρος Επιτροπής, ο κύριος Γιούγκα, μας υποσχέθηκε ότι θα πλουστεύσει τη γραφειοκρατία και σήμερα είδαμε ότι θα συμβεί το αντίθετο. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα ότι η πρόταση αυτή κατ' ουσίαν είναι απάτη, διότι μας λένε ότι τα κράτη-μέλη που δεν επιτιμούν τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς μπορούν να εξαιρεθούν. Αυτό όμως μόνο εφόσον τηρούνται αυστηρά τρία κριτήρια ε, τα οποία ε, όλα είναι προσβλητά. Δηλαδή αυτό που προτείνεται είναι το ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να κρυφτούν πίσω από μία απόφαση στην ευρωπαϊκή αγορά θα επιτρέπονται αυτοί οι οργανισμοί και εκ των υστέρων ε, τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει μόνα τους να βρουν μια λύση έναντι αυτών των οργανισμών. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι λάθος και έναντι των κρατών και έναντι των πολιτών. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω να ακουστούν αυτά τα λόγια, να μεταφερθούν στον Επίτροπο και νομίζω ότι ε, τα άκουσα έτσι και σήμερα στην Επιτροπή ΕΝΒΗ. Πολύ ωραία. Η κυρία Μακίνες έχει το λόγο. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, οποιαδήποτε και να είναι η άποψή μα για το ζήτημα αυτό, νομίζω ήταν εξαιρετική η παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα είπε ξεκάθαρα ότι εξαρτώμεθα απολύτω από την γενετικά τροποποιημένη σόγια ω πηγή πρωτενη. Οποιαδήποτε λοιπόν πρόταση λέει ότι μία νυχτή θα αλλάξουν τα πράγματα δεν είναι σωστή, είναι ανεδαφική. Υπάρχει εδώ πέρα ένα συγκεκριμένο δίλημα όμως. Έχουμε μία πολιτική πρόταση ευφυή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει ότι τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια. Η δική μας τώρα επιτροπή δεν συμφωνεί βέβαια για τα πάντα, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει γενικότερη συνένεση για την πρόταση αυτή. Αλλά μάλλον δεν θέλουμε την ίδια συνέχεια όσον αφορά την έκθεση αυτή. Άλλα πράγματα θέλουμε να δούμε στο μέλλον. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι η πρόταση θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να απαγορεύσουν τη χρήση, αλλά όχι την κυκλοφορία την εισαγωγή μεταλλαγμένης σόγιας. Για ποιο λόγο να την εισάγει όμως κανείς αν δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει. Αυτό το καταλαβαίνω. Επίσης αναφερθήκατε στις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, σε μια ανάλυση κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο περισσότερα στοιχεία γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Δεκάστρο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρο. Όντως πολλά πράγματα ήδη υπόθηκαν. Σίγουρα, όπως το ακούσατε, η δική μου πολιτική ομάδα είναι επιφυλακτική και θέλουμε να ακολουθήσουμε την πρόταση του εισηγητή Ντες. Αναμφίβολα η πρόταση αυτή που υπέβαλε ο Επίτροπος κατά κάποιο τρόπο προκαλεί αυτή τη στιγμή μια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη μας ότι το 95% των ε, αναγκών μας σε σόγια είναι σόγια η οποία εισάγεται και είναι κυρίως μεταλλαγμένη σόγια. Μόνο και μόνο αυτό ως δεδομένο ξεκινά μια ολόκληρη συζήτηση. Δεν μπορούμε τώρα να δείξουμε υποκρισία, δηλαδή από τη μία πλευρά να λέμε ότι είμαστε κατά των γενετικά ανθρωποποιημένων οργανισμών και από την άλλη να συνειδητοποιούμε ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα χωρίς ε, αυτούς τους 37 εκατομμύρια τόνους που εισάγουμε. Προκαλείται λοιπόν μια γενικότερη συζήτηση και νομίζω ότι σε τελική ανάλυση περισσότεροι θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει την πρόταση αυτή. Μέχρι να γίνει όμως αυτό θα έχουμε κάπως απο, αποσαφηνίσει τα πράγματα. Ενδεχομένως να καταφέρουμε να δώσουμε κάποιες συγκεκριμένες ενδείξεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την άλλη ενδεχομένως να καταφέρουμε να αφουγκραστούμε καλύτερα και τις ίδιες ανησυχίες των καλλιεργητών, των γεωργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν υπάρχουν πολλά να προσθεθούν σε αυτά που ήδη ελέγχθησαν. Ισχύει το εξής, ε, ήδη σήμερα υπάρχουν χώρες και η δική μου η περιοχή όπου οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, μπορούν να παρετηθούν από τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, τροφίμων, ζωοτροφών. Και αυτό το λένε με ετικέτες ε, στα προϊόντα τους. Και εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτή είναι μια απόφαση δική τους που μπορούν να τη λάβουν, κανένα πρόβλημα. Η πρόταση λοιπόν ε, για μένα, ξέρετε, πρέπει να σας πω ότι είναι λιγάκι περίεργη. Ε, διαβάζω την πρόταση και διαβάζω ότι όλα αυτά ε, δεν θα επηρεάσουν την κοινή αγορά. Αλλά τι να πω τώρα, μεγαλύτερη στρέβλωση ανταγωνισμού δεν υπάρχει. Για σκεφτείτε τι θα γίνει στην χειροτροφία εάν σε μία χώρα επιτρέπονται οι γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και στην άλλη όχι. Προφανώς και εδώ μιλάμε για στρέβλωση ανταγωνισμού. Όπως είπε και η κυρία Μακίνες, αν αυτό ε, έγινε με τη μορφή προβοκάτσια, τότε ήταν πραγματικά μία πολύ επιτυχημένη προβοκάτσια. Πριν από δύο εβδομάδες ο Επίτροπος ε, θέλησε να τα υπερασπιστεί όλα αυτά και πραγματικά έκτοτε ανησυχώ κι εγώ όσον αφορά στις αρμοδιότητες των άμεσα εμπλεκόμενων. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι με όλη αυτή τη συζήτηση διαπιστώνουμε πόσο υποκριτική είναι η συζήτηση για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Αρχίσαμε να συζητάμε για αυτούς, ε, παραπέμψαμε το θέμα στην αρμοδιότητα των κρατών μελών ε, και τώρα σιγά σιγά στην Ευρώπη ε, υποτίθεται έχουμε μόνο κάποια εκτάρια που καλλιεργούνται στην Ισπανία και τίποτα άλλο. Δηλαδή τι γίνεται, συζητάμε για πράγματα που δεν υπάρχουν. Το βασικότερο θέμα είναι οι εισαγωγές, οι και η χρήση ε, των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να τα σκεφτούμε όλα αυτά και όσον αφορά και την ε, χρήση πρωτεϊνών στην Ευρώπη. Πάντως ε, αυτή η πρόταση της Κομισιόν δεν μας βοηθάει να προχωρήσουμε, είναι σαφώς ένα βήμα προς τα πίσω. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι λοιπόν ακούσαμε όλους τους ερωτώντες. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι προσδοκίες μας ε, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δυστυχώς το πρόβλημα θα παραμείνει ακόμα και αν αναπέμψουμε αυτήν την πρόταση. Παρόλα αυτά θα πρέπει να ξαναγίνουν σοβαρές συζητήσεις για αυτό το θέμα. Αλλιώς, αν δεν γίνουν σοβαρές συζητήσεις, δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά. Δεν ξέρω αν εμείς μπορούμε να αποφασίσουμε το τι θα γίνει στην παγκόσμια αγορά. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Νίκο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους βουλευτές για τα σχόλια και τις ερωτήσεις τους. Θα προσπαθήσω να ενοποιήσω κάποια ερωτήματα. Ιδίω αυτό το οποίο επανήλθαν συζήτηση αρκετέ φορέ. Πρώτα απ' όλα, πολλέ φορέ ετέθη το ζήτημα τη ενιαία αγορά και τις δυνητικές ανάγκες ελέγχου συνόρων, κατοφλήν κτλ. Θέλω να σας πω ότι είναι προφανές πως όταν μιλάμε για απαγόρευση της χρήσης στην επικράτεια ή σε ένα συγκεκριμένο μέρος, σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια, δεν μιλάμε για την απαγόρευση μετακίνησης ε, στα επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα η συνοριακή ελληνική δεν είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτό αναλύθηκε το ζήτημα της νέας αγοράς εντελεχέστατα και το ισχύον και εκτιμένο προβλέπει τις προποθέσεις υπό τις οποίες έχουμε ε, το άρθρο 36 συγκεκριμένα που δίνει δυνατότητα στα κράτη-μέλη να παρεκκλίνουν από τους κανόνες της ενίας αγοράς δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε τελευταία παρέκκληση που χρησιμοποιείται και σε πολλού άλλου τομεί μάλιστα μεταξύ αυτών και στον τομέα της γεωργίας. Νομίζω το ξέρετε άλλωστε πολύ καλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα άλλο θέμα είναι κατά πόσον είναι δυνατή η παραγωγή περισσότερων πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Πρέπει να σας πω ότι πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή κατά 20 φορές. Υπάρχει χώρος στην Ευρώπη. Μόνο αν σταματήσουν να καλλιεργούνται άλλα είδη μπορούμε να αυξήσουμε το ποσοστό των, της των πρωτεϊνών. Και βέβαια να λάβουμε υπόψη και τις ε, φυσικές και κλιματικές συνθήκες για την προστασία αυτών των ε, καλλιεργειών. Ακόμη και αν ήταν ε, τα εδάφη άδεια θα μπορούσε να καλυφθεί η ανάγκη για τις πρωτεΐνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν το συζητήσαμε, και επανέρχομαι στην νέα αγορά, σας υπενθυμίζω ότι στο υφιστάμενο σύστημα μπορεί κανείς να ενεργοποιήσει τη ρήτρα διασφάλισης που χρησιμοποιήθηκε μάλιστα από αρκετά κράτη-μέλη κατά το παρελθόν. Αυτό έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το προτινόμενο μέτρο. Γιατί ορισμένα εδάφη εξαιρούνται τη έννοια αγορά για την περίοδο ισχύω τη ρήτρα διασφάλιση. Πολλέ φορέ έχει γίνει επίκληση τη ρήτρα και δεν δημιουργήθηκε κανένα από τα προβλήματα που αναφέρονται στη σημερινή συζήτηση. Νομίζω λοιπόν ότι ήδη έχουμε την εμπειρία μα και η μόνη διαφορά είναι ότι με τη ρήτρα διασφάλιση, η επίκληση αυτή τη ρήτρα, συνδέεται ή σχετίζεται με νέα επιστημονικά στοιχεία, ενώ εμείς χρησιμοποιούμε ως λόγο άλλους θεμητούς παράγοντες. Αλλά η ίδια επίπτωση θα είναι για την αγορά. Η ΕΦΣΑ αναφέρθηκε πολλές φορές. Πολύ ξεκάθαρα θέλω να πω ότι ήταν απόφαση του Ευρωπαϊκού Συστήματος να υπάρχει μία και μόνη επιστημονική αρχή που θα παίρνει αποφάσει για τα ζητήματα ασφάλεια τροφίμων. Δεν θα πρέπει να κατηγορούμε την ΕΦΣΑ που δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τη θεμελιώδη αντίθεση που εξέφρασαν αρκετοί από εσά ε, στι γενετικέ μεταλλάξει. Δεν μπορώ να αποδοθώ στην επιστήμη, αλλά αφήνονται σε άλλου θεμητού παράγοντε, ηθικοί ε, παράγοντε, ε, πολιτισμικοί παράγοντε κτλ. Ο ρόλο τη ΕΦΣΑ είναι άλλο. Είναι να κάνει επιστημονικέ εκτιμήσει. Και όπω είπε και η κυρία Αγιούσο, και εγώ είμαι πεπισμένος ότι αυτό γίνεται με βάση τα ανώτατα δυνατά επιστημονικά πρότυπα. Αν τώρα είναι θετικό το αποτέλεσμα και δεν έχει όμω αποτέλεσμα ψηφοφορία από το Συμβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει η Επιτροπή να αποφασίσει με βάση τα επιστημονικά στοιχεία και δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ακολουθούμε στις αποφάσεις μας τις επιστημονικές μαρτύρες, τα επιστημονικά στοιχεία. Σε σύγκριση με την σημερινή κατάσταση προσφέρουμε μια επιλογή για τα κράτη-μέλη που έχουν θεμελιώδεις άλλους δηλαδή θεμητούς παράγοντες να προβούν σε αυτή την αυτοεξαίρεση, στο opt-out. Νομίζω ότι θα πρέπει να συγκρίνουμε την κατάσταση όσο έχει τώρα με την κατάσταση που προτείνουμε και να μην έχουμε στο μυαλό μας ε, μια ιδεατή κατάσταση. Γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Ένα πολύ σημαντικό ερώτημα της κυρίας Μακίνες αφορούσε το κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο. Θα το απαντήσω και αυτό. Πράγματι, αν η απαγόρευση ίσχυε για όλη την επικράτη της Ένωσης, δεν θα είχε νόημα να γίνονται εισαγωγές. Όμως, εάν έχουν λίγα επιλεγμένα εδάφη, τα οποία θα, θα εξαιρεθούν και πάλι θα πρέπει να είναι δυνατόν να υπάρξει αγωγή πρωτεϊνών μεταλλαγμένων για ζωοτροφές για παράδειγμα. Να μεταφερθούν εντό Ένωση και να καταλήξουν στο σημείο όπου θα χρησιμοποιηθούν. Μπορούμε να αφήσουμε ανοιχτή αυτή τη ε, δυνατότητα και μάλιστα πρέπει να το εξασφαλίσουμε κιόλας γιατί τέλος φτάνουμε στο πρόβλημα των συνοριακών ελέγχων που δεν είναι πρόθεσή μας. Κοινωνικο-οικονομικός αντίκτυπος τώρα σημαντικότατο ζήτημα. Είπα όμως και στην εισαγωγική μου ομιλία ότι μπορεί να εκτιμηθεί με εξόπιστο τρόπο μόνο εφόσον είναι γνωστό σε ποιο βαθμό θα απαγορευτεί η χρήση και σε ποια εδάφη. Ιδάλλως έχουμε μια εκατομμύρια επιλογές που δεν είναι δυνατόν να τις αναλύσουμε σοβαρά. Άρα, άρα τα κράτη-μέλη είναι αυτά που πρέπει να αποφασίσουν εν τέλει. Αν μπορούν να ακολουθήσουν το opt-out και να αναλύσουν, όπως είπα, τον κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο. κύριος Κάστρο είπε ότι δεν θα πρέπει να είμαστε υποκριτές στη συζήτηση αυτή. Είναι ένα θέμα αυτό. Γιατί πρέπει να είναι σαφές ότι σήμερα η κατάσταση πώς έχει. Τα κράτη-μέλη ψηφίζουν κατά ή απέχουν από την ψηφοφορία στην Ευρωπαϊκή Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων. Δεύτερον, χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό μεταλλαγμένες ζωοτροφές, ενώ κατηγορούν μετά την Κομισιόν που εγκρίνει τα μεταλλαγμένα αυτά προϊόντα. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν αυτή την κατάσταση να το αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Άρα νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και να πούμε ότι πάντοτε υπάρχει επιλογή. Παραλαμβάνω, σήμερα είναι επιλογή το να ψηφίσει κάποιος κατά. Αν υπήρχε πλειοψηφία κατά, καταψηφιζόταν και τέλειωνε το θέμα. Δεν υπάρχει όμως το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει ψήφος. Και αν δεν αλλάξει, θα έχουμε δύο γύρους προφοριών και στην επιλογή, στην Επιτροπή Συγγνώμη Εφέσεων ή Προσφυγών μετά. Και έχουμε ένα τρίτο υπέρ, ένα τρίτο κατά, ένα τρίτο αποχή. Όλοι, για να μην πω τέλο πάντων, πολύ σιωπηρά περιμένουν να εγκριθεί γιατί πρέπει να το χρησιμοποιήσουν στο σπίτι τους, στη χώρα τους, αλλά κατηγορούν μετά την Κομισιόν. Εμείς είπαμε να δώσουμε μια πραγματική νόμιμη επιλογή σε αυτούς που είναι κατά για να αυτοεξαιρεθούν και να δούμε ποια είναι η κατάσταση στην Ευρώπη. Το σημαντικό είναι και ναι, το παρατήρησα και εδώ και στην Επιτροπή Έμβη. Η ομοφωνία στην άρνηση. Κάτι που είναι σπάνιο. Είστε όλοι κατά εδώ. Αλλά πρέπει να πω ότι είναι σημαντικό να αναλύσουμε γιατί είναι ο κόσμος αντίθετος αυτή την πρόταση. Για δύο βασικούς λόγους. Υπάρχει μια κατηγορία που είναι κατά των μεταλλαγμένων και έχουν διαφορετικούς λόγους απέναντι σε αυτούς που είναι υπέρ. Προσπαθούμε εμείς να βρούμε με ποιο τρόπο θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση περισσότερο για την ψηφοφορία επί της έγκρισης των μεταλλαγμένων στο μέλλον. Εμείς πρέπει να σας πω, πανεξετάσαμε και αναλύσαμε όλες τις θεωρητικές και τεχνικώς εφικτές επιλογές μπορείς να κάνει να φανταστεί σε αυτή την κατάσταση. Και καταλήξαμε μόνο σε αυτή τη λύση, είναι η μόνη που μπορεί να λειτουργήσει, γιατί με άλλες θα μιλούσαμε είτε για κατάργηση ε, συνθήκης, η επαναδιαπραγμάτευση, η αλλαγή μηχανισμών ψηφοφορίας κτλ. Δεν θα το στηρίζατε κάτι τέτοιο, είμαι απόλυτα βέβαιος. Επομένως, το θέμα είναι ότι ε, αν θέλουμε να αλλάξει κατάσταση, αυτή είναι η λύση. Και αυτή τη λύση προτείνουμε. Εσείς έχετε βέβαια κάθε δικαίωμα να την εξτάσετε και να την απορρίψετε. Τότε όμως ξαναγυρίζουμε στην κατάσταση που έχουμε τώρα και δεν υπάρχουν πολλές άλλες επιλογές να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να στο λόγο στον κύριο Ντές ε, και δεν σας ζηλεύω κύριο Ντές, πρέπει να σας το πω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαρίστω ε, αναλαμβάνω αυτό το καθήκον, μου κάνει μεγάλη χαρά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναντέλφους που έλαβαν το λόγο. Ε, θέλω να τα υπογραμμίσω όλα αυτά που ελέγξαν. Δεν ξέρω τι έχω να επικρίνω. Αυτά που είπε η Αυστριακή συνάδελφη τα στηρίζω ανεπιφύλακτα. Ε, παρότι ο κύριος Γιούγκερ έχετε από τη δική μου την πολιτική οικογένεια, εδώ παίζει ένα άσχημο παιχνίδι και εμείς δεν θα το δεχτούμε. Το θέμα αυτό δεν ενδείκνυται για παιχνίδια, δεν είναι θέμα που μπορεί ε, να είναι αντικείμενο αντιπαράθεση ανάμεσα στους θεσμούς. Κύριε Νίκο, ε, θέλω να σας ε, συγχαρώ. Είσαστε πιστός υπηρέτης του αφεντικού σας ε, και εάν ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίες ή εργαζόσασταν στην ελεύθερη αγορά θα σας έλεγα ότι είστε ο καλύτερος πολιτής. Μπορείτε να πουλήσετε ένα σαραβαλάκι για αυτοκίνητο της χρονιάς. Εμείς όμως το σαραβαλάκι αυτοκίνητο δεν θα το αγοράσουμε, θα το στείλουμε πίσω. Γιατί αυτό το σαραβαλάκι δεν ενδείκνεται να φέρει κάτι νέο και καλό στην Ευρώπη. Ελπίζω λοιπόν να βρούμε την απαραίτητη πλειοψηφία για να κλείσει το θέμα χωρίς πολλές ε, συζητήσεις. Ο κύριος ε, Τζοβάνι Λαβία που είναι αρμόδιος ε, στην Επιτροπή ΕΝΒΗ έχει την ίδια απόψη με εμάς. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν αντίθετα από αυτά που πιστεύει η Επιτροπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε ούτε όμως και καινούργιο αυτοκίνητο θα μας δώσετε ή θα αποκτήσουμε ούτε θα αγοράσουμε και το παλιό. Μέχρι 15 και 16 Ιουλίου η κατάσταση τροπολογιών. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Το θέμα είναι πολύ λεπτό και είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί η καλύτερη λύση. Σας παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ αύριο να έρθετε με τις ε, κάρτες σας διότι, διότι αύριο θα ξεκινήσουμε με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Μην ξεχάσετε να καλέσετε τον κύριο Νίκολσον. Ε, το θέμα είναι πολύ δύσκολο. Πρόκειται για την παραγωγή αυγών. Για το TTIP, για το γαλακτοκομικό τομέα, κόπα κοσέκα. Κάτω λοιπόν στο σαλόνι. γι' αυτά θα κουβεντιάσουμε. Ευχαριστώ πολύ.